Guten Morgen, liebe Μέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάει στον Καναδά και με την ICAO, ICAO συζητήσαμε θέματα ασφάλειας των αεροπορικών μεταφορών και μετά σε σχέση με συζητήσεις μάθαμε ότι στην Αίγυπτο η πτήση Α320 από το Παρίσι προς Κάιρο είχε συντριβεί και 66 θύματα ήταν το αποτέλεσμα αυτής της ε, συντριβής. Θέλω να υπενθυμίσω φυσικά ότι τα συλληπιτήριά, μου, συλληπιτήριά μας ε, προς την οικο, τις των θυμάτων. Ένα λεπτό θα αποτίσουμε φόρο τιμής παρακαλώ στα θύματα. Vielen Dank. Σας ευχαριστώ πολύ. Zunächst mal haben Sie... Πρώτα Herr όλα Έχουμε τις αποφάσεις, έχετε τις αποφάσεις από χθε ε, το βράδυ των συντονιστών. Αν δεν υπάρξουν κάποιες αντιρρήσεις μέχρι το μεσημέρι 12.30 ώρα, θα θεωρηθεί ότι κυρώνονται και εγκρίνονται. Και περνάμε έτσι αμέσως στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης για τον κανονισμό για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Αεροπορίας. Όπως όλοι θα θυμόσαστε, η Επίτροπος Μπούλσα είχε παρουσιάσει το Δεκέμβριο το πακέτο μέτρων, τη δέσμη μέτρων για την ε, ε, υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Ασφάλειας Αεροπορίας. Ο εισηγητής μας ε, Μαριαν Γιάννου Μαρινέσκου εξεπώνησε την έκθεσή του στη συνέχεια. Στην αρχή έχουμε και όλα αρκετούς προσκεκλημένους για τα θέματα των μη επανδρομένων αεροσκαφών Πρόκειται για τον κύριο Μπέργεν από την European Cockpit Association, Ούκαλα από την Φινλανδική Οργάνωση και τον κύριο Τούμελ από την Γαλλική EJC. Ερικ Σιβέλ που δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε λόγω ε, υγείας, λόγω, λόγω υγείας να παραστεί. Δεν ήταν δυνατόν να προσκαλέσουμε άλλον επαΐοντα όμως ο Λουτσίγετ από πλευράς ε, της οργάνωσής του είπε ότι ε, μπορεί να συνεργαστεί και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους επαΐοντες εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Καλώς ήρθατε θερμά και εύχομαι να έχουμε θετικές συζητήσεις επί των θεμάτων αυτών. Ο κύριος εισηγητής Μαριάν Γιάν Μαρινές που θα λάβει τον λόγο μετά η προσκεκλημένη μας. Thank you, ε, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία, του Σκιώδης. Είχαμε ήδη μια συνάντηση και θα έχουμε άλλη μία σε δύο εβδομάδες. Σε γενικές γραμμές ε, είναι μια καλή πρόταση της Επιτροπής και νομίζω προς το συμφέρον των δραστηριοτήτων της ΕΑΣΑ των γενικών δραστηριοτήτων και κάποιων ειδικών τις οποίες εκπληρώνει αυτή τη στιγμή ο οργανισμός. Θα πω απλώς ε, δύο λόγια σχετικά με κάποιες καινούργιες διατάξεις στον κανονισμό Είμαι υπέρ της ε, συμμετοχής της ε, στα θέματα ασφαλείας, αλλά μόνο στα θέματα ασφαλείας που έχουν σχέση κυρίως με τον κυβερνοχώρο, εξοπλισμό αερολιμένων που έχουν σχέση με θέματα ασφαλείας, επίσης για θέματα εκπομπών περιβαλλοντικά, και άλλοι φορείς θα συμμετάσχουν, αλλά δεδομένου των διατάξεων των παραρτημάτων της ΙΚΑΟ, σχετικά με την πιστοποίηση του εξοπλισμού εδάφους και του προσωπικού εδάφους, νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα προς τα εμπρός γιατί θα ενέχει πλεονεκτήματα για τις ε, δραστηριότητες αυτές των αερολιμένων, για τα του προϋπολογισμού, για ένα μέρος του άχθους και μέρος των ε, καθηκόντων της Eurocontrol και αυτό νομίζω ότι θα είναι θετικό για τον οργανισμό. Τώρα, για τις ε, ζώνες συγκρούσεων και για την συνεχή καταγραφή των δεδομένων πτήσης, real time, δηλαδή διαβίβαση προς το έδαφος ώστε να είναι αυτά διαθέσιμα σε συνεχή χρόνο, σε περίπτωση ατυχημάτων, Γενικώ είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον, για την ασφάλεια των πτήσεων και των αερομεταφορών. Εξού και πρότεινα αυτή την εκδήλωση σήμερα. Θα πρέπει νομίζω να εγγραφεί στον κανονισμό, να μην περιμένουμε μόνο τις ε, κατεξόδοτης πράξεις της Κομισιόν, θα πρέπει να αποφασίσουμε κάποιες ε, γενικές γραμμές, ταυτοποίηση, καταχώρηση, geofencing. Κάποια στοιχεία θα πρέπει να ενσωματωθούν στον κανονισμό και γι' αυτό ήθελα να ακούσω και την άποψη των εμπειρογνωμόνων. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρώτος θα λάβει τώρα τον λόγο ο κύριος Τόμας Μπίλτενμπέργκερ από την European Cockpit Association. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητέ εισηγητά, αγαπητοί ευρωβουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας προσφέρατε να σας παράσχουμε την πραγματογνωμοσύνη μας. αναφέρομαι ειδικά στα μη επανδρομένα αεροσκάφη όταν ένα, ε, ε, πετά σε ένα ε, διεθνές δίκτυο για μια γερμανική εταιρεία, είμαι πρόεδρος της εταιρείας European Cockpit Association των πιλότων και είμαι και μέλος του Συμβουλίου της ICAO στο Μόντρεαλ. Μια και πιέζει ο χρόνος, θα επικεντρωθώ σε τρία κύρια θέματα που θεωρώ ότι είναι σημαντικά για μια ασφαλή λειτουργία μη επανδρομένων αεροσκαφών το, στους εθέρες. Πρώτον, η εφαρμογή και η συμμόρφωση με τους κανόνες και κανονισμούς. Δεύτερον, η ανάγκη να υπάρχουν άδειες για τέτοιες πτήσεις και τρίτον τεχνική περιορισμοί για την χρήση τέτοιων μη επανδρομένων αεροσκαφών. Χτυπούν στην πόρτα μας τα μη επανδρομένα αεροπλάνα και θα παραμείνουν. Πολλές φορές όμως ε, γίνονται αυτές οι πτήσεις ε, με μη επαρκείς κανόνες η ασφαλής λειτουργία των μη επανδρομένων αεροσκαφών είναι προ όφελο όλων, του κοινού, των ρυθμιστικών αρχών και φυσικά και τη ίδιας της βιομηχανίας αεροσκαφών, μη επανδρομένων αεροσκαφών. Υπάρχουν σημαντικά μελήματα που πρέπει να τεθούν όταν αναφερόμαστε σε κανονισμούς ε, με βάση τους κινδύνου με μια νέα μεθοδολογία, σε ένα ε, ανεξερεύνητο τομέα των ε, δράσεων στου εθέρες όπω είναι τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι κύριες ανησυχίες μας αφορούν την ανοιχτή κατηγορία των μη επανδρομένων αεροσκαφών, open category. Υποτίθεται ότι έχουν χαμηλό κίνδυνο, χαμηλό επίπεδο κινδύνων και είναι, ε, λειτουργούν χωρίς ε, εποπτεία των ε, ε, αεροναυτικών αρχών. Και Υπάρχει εδώ ε, και το θέμα του, του σκυροδέματος που ε, αντίστοιχου βάρου σκυροδέματος αυτών των ε, αεροσκαφών. Πρέπει να δούμε το θέμα των, από, της απογείωσης και προσγείωσης αεροσκαφών, στρατιωτικών και μη και όλα αυτά σε 150 μέτρα από το έδαφος. Μια και οι εθέλες είναι ενιαίοι, το να πετούν όλοι σε, ένα, σε μια περιοχή θα πρέπει να συνεπάγεται να συμμορφώνονται με τις ίδιες αρχές, αν όχι και με τους ίδιους κανόνες και κανονισμούς. Ταυτόχρονα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν ε, ενδιαφέρονται καν πολλοί από αυτούς ε, που κάνουν τέτοιες πτήσεις ε, στο να σεβαστούν τέτοιους κανόνες. Και όσον αφορά τις ε, συναντήσεις ε, με, ε, πολιτική, με αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας δείχνουν αυτές οι καταστάσεις ότι δεν έχουν καν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που προκαλούν οι πτήσεις τους. Θα έρθω σε τρία σημεία που θέλω να αναφέρω. Πρώτον, αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και κανονισμών. Υποχρεωτική καταχώρηση σε μητρώα αυτών των αεροσκαφών ώστε να μπορούν να ταυτοποιούνται οι πτήσεις τους. Αν δεν μπορούν όμως να εφαρμοστούν και να είναι σεβαστοί οι κανόνες δεν θα έχει νόημα η υπόθεση. Ελπίζουμε ότι θα είναι δυνατόν να, να ε, ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Κάποιες εθνικές αστυνομικές αρχές είναι πολύ χλιαρές στο να αναλάβουν επιπρόσθετες αρμοδιότητες και ευθύνες με ένα τέτοιο τομέα που θα υποπτεύουν. Δεύτερο, κάθε πιλότος τέτοιων αεροσκαφών πρέπει να έχει άδεια πτυχίο που θα αναφέρεται αναλογικά στους κινδύνους τέτοιων πτήσεων και που θα εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. Μόνο τα παιχνίδια εντός εισαγωγικών που δεν δημιουργούν οποιαδήποτε προβλήματα θα μπορούν να εξαιρούνται τα παιχνίδια από τέτοιου είδους κανόνες και κανονισμούς. Με ένα συγκεκριμένο βάρος για παράδειγμα μέχρι ενός συγκεκριμένου βάρους κτλ. Και τότε θα μπορούσαν να υπάρχουν πιο χαλαροί κανόνες. Όταν θα υπάρχει και πραγματικά πραγματογνωμοσύνη επιστημονική που θα δείχνει ότι για τις ανώτερες κατηγορίες θα μπορεί να υπάρχει ειδική αντιμετώπιση. Τρίτη παρατηρήσή μου είναι η τεχνική περιορισμοί όσον αφορά τη λειτουργία τους. Θα πρέπει να είναι αναγκαίο να υπάρχει αντιστάθμιση για το ότι δεν θα υπάρχει ε, επί ε, του αεροσκάφους επιλότος. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει, δεν είναι, δεν θα πρέπει να είναι ικανό ένα τέτοιο αεροσκάφος να εγκαταλείψει την ε, περιοχή στην οποία θα επιτρέπεται να κινείται και δεν θα επιτρέπεται να έχει μεγαλύτερη ακτίνα δράσης από εκείνη που θα επιτρέπεται. Και αν θα επιτρέπεται να γίνεται κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να αποφεύγει τις ε, συγκρούσεις ή επαφές με άλλα αεροσκάφη που θα πετούν σε αυτές τις περιοχές avoidance, αυτόματη αποφυγή δηλαδή, αυτόματη αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και κανονισμών, υποχρεωτική καταγραφή, άδειε για πιλότου, τεχνική περιορισμή για τα αεροσκάφη. Είναι απόλυτα αναγκαίοι κανόνε. Οι κανόνε και οι κανονισμοί για να πετύχουμε αυτή την κατάσταση πραγμάτων είναι αναγκαίοι για να μην καταλήξουμε σε ένα χάο στου εθέρε μα. Είναι λοιπόν ευθύνη των νομοθετών να το επιτύχουν. Αυτό σα ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας εκθέσατε. Γιάκου Ανούλα τώρα, από την Φινλανδική Αρχή. Έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Σιγητά, αγαπητέ Ευρωβουλευτές. Έχουμε μια μοναδική δυνατότητα να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρώπη. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που κινούνται ε, στην ίδια περιοχή, στα ίδια, σίγουρα χρειάζονται και οι ίδιοι κανόνες, ε, δίκτυα ασφαλείας κτλ. Και είχαμε πει και με τη ΔΟΠΑ ότι πάντοτε ε, έπρεπε να λαμβάνουμε υπόψη αυτό, γιατί σίγουρα θα έχουμε στο κοντινό μέλλον αυτές τις εξελίξεις. Είναι πολύ μικρότερα τα αεροσκάφη για τα οποία χρειάζεται νέα σκέψη, καλύτεροι κανόνες. Οι εταιρείε σε αυτόν τον τομέα συχνά είναι μικρές ε, νεοσυσταθήσεις εταιρείε. Και θα πρέπει να τους δώσουμε τη δυνατότητα να επιτύχουν. Δεν μπορούμε να τις φορτώσουμε με αχρίαστο κόστος ε, και διοικητικό βάρος που μάλιστα θα έχει και πολύ περιορισμένη προσθέμενη εξέσωτη την ασφάλεια. Οι κανόνες επίσης ε, θα πρέπει να βασίζονται στις επιδόσεις. Ε, η τεχνολογία αναπτύσσεται με ταχύτητους ρυθμούς ε, και οι τεχνικές απαιτήσεις πολύ γρήγορα καθίστανται απαρχιωμένες. Για παράδειγμα, στο φιλανδικό κανονισμό εστιάζουμε στην έκβαση και το επίπεδο ασφάλειας που πρέπει να επιτευχθεί. Αλλά δεν λέμε πώς οι operators, οι φορείς θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν το, το πώς. Επίσης, ε, εφαρμόζουμε νέους εφαρμοστικούς κανόνες. Χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες ε, ε, Open Specific Certified τις επιχειρήσεις. Το ένα, το τρίτο θα εντάσσεται στην... Μάλλον μοιάζει πολύ με τα όσα ισχύουν για τα επανδρομένα αεροσκάφη. Στη δεύτερη περίπτωση χρειάζεται και η συμβολή των εθνικών αρχών. Και έπειτα υπάρχει αυτή η ανοιχτή κατηγορία, το open category, που νομίζω θα μπορούσε να γίνει πολύ περιοριστική. Ιδίω αν ληφθούν υπόψη αρχικέ ιδέε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην έχουμε λοιπόν τον διοικητικό άχθο σε αυτή την κατηγορία, την ανοιχτή κατηγορία, θα πρέπει να βασίζονται στον κίνδυνο και σε επιδόσει ε, οι διατάξει και να αφήσουμε περιθώρια λοιπόν στα κράτη-μέλη είναι σαφές ότι στις άλλες δύο κατηγορίες χρειάζεται ένας ενίος ευρωπαϊκός κανονισμός για να υπάρχει ανταγωνισμός και ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και στην open κατηγορία χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Επαρκεί πιστεύω ένα υψηλό επίπεδο και θα επιτρέψει στον κλάδο να θεσπίσει κάποια πρόταση. Υπάρχουν διάφορα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Οι μηχανικοί οποίοι παίρνουν κάποιε ε, αεροφωτογραφίε, ε, μεσίτε, κτηματομεσίτε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι διαφορετικέ αυτέ ε, δραστηριότητε και να μην περιπλέξουμε το έργο όλων αυτών των φορέων. Θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο επίση την πρόθεση τη ασφάλεια, ίσω να έχουμε κάποιε κινητέ εφαρμογέ για να μπορούν να καταλάβουν αυτοί που μπορούν ή δεν μπορούν να, να πετούν υλικό καθοδήγηση στα 150 μέτρα που είναι και το κατώτατο όριο για τις απανδρομένες πτήσεις και τα λοιπά πρέπει να ληφθεί υπόψη. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες πτήσεις κάτω από τα 150 μέτρα που κυρίως είναι στρατιωτικές πτήσεις της ελικοπτέρων. Σε αυτή κατηγορία η απαιτούμενη εμπειρογνωμοσύνη πρέπει να αναζητηθεί σε εθνικό επίπεδο. Τα προβλήματα τη ανοιχτή κατηγορία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε παρκώ σε ενωσιακό επίπεδο. Ή αν μπορούσαμε, θα είχαμε ε, πολύ περιοριστικού κανόνε σε πολλέ περιπτώσει. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλη πρόκληση να βρούμε ε, την ισορροπία μεταξύ του επίπεδου ασφαλεία ε, και περιθωρίων. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα μία επανδρομένα, πούμε ότι πετούν σε κάποια σε κάποια περιοχή που, δεν, που ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και χρειάζονται και κάποια αντίμετρα. Καλό θα είναι υπάρχει ένα σύστημα εντοπισμού αναγνώρισης και όταν ισχύουν, όταν υπάρχουν αυτά τα συστήματα, τα μη ε, αναγνωρισμένα ε, αεροσκάφη θα μπορούν να θεωρούνται απειλή. UTM χρειάζεται. UAS Traffic Management θα πει αυτό. Είναι κάτι που ίσως δεν το χρειαζόμαστε ακόμη με τον όγκο που έχουμε τώρα στην ενεργοκυκλοφορία, αλλά αν το αναπτύξουμε σίγουρα χρειάζεται κάποιο χρόνο για να είναι έτοιμο και θα περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία για να βελτιώσει την ασφάλεια. Υπήρξαν πάρα πολλά συμβάντα μεταξύ πανδρομών και μη επανδρομένων σε χώρες που έχουν δυσκύνει τους κανονισμούς. Τους μικρούς φορείς ε, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να του δώσουμε περισσότερε πληροφορίε, να του δώσουμε τα εργαλεία για να καταλάβουν ε, τη δομή του εναέριου χώρου κτλ. Και έτσι θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί, όχι τόσο με έναν πολύ αναλυτικό κανονισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αζημέρ τώρα από τον Γαλλικό Οργανισμό έχει τον λόγο. Dear Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής, ευχαριστώ τον εισηγητή για την ευκαιρία αυτή για να μοιραστούμε την ευκαιρία μας μαζί σας. Οι κανονισμοί αυτοί δημιουργήθηκαν το 2012 και επικαιροποιήθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο κλάδος αναγνωρίζει ότι ο κανονισμός αποτυπώνει την ταχύτατη ανάπτυξη της αγοράς. 1.800 φορείς υπήρχαν περίπου στα μέσα του 2015, ε, μισή εκ των οποίων στα διαφημιστικά, ένα πέμπτο στις κατασκευές. Ε, πρόκειται για μια ταχαίως αναψιόμενη αγορά. the development of the industry. Ε, πέρυσι συναισθήθη ένας φορέας που εκπροσωπεί τους φορείς του κλάδου και συζητεί επίσης τεχνικά θέματα και θέματα ασφαλείας όπως και την προώθηση της όλης βιομηχανίας. Ως παράδειγμα της δουλειά που γίνεται, στις πρώτες δύο συναντήσεις δημιουργήθηκε μια task force για να παράσχει τεχνικές λύσεις μέσω και μακροπρόθεσμα για τις ε, πτήσεις ε, μεγάλης διαρκείας και επί τη βάση της, της εμπειρίας αυτής θα ήθελα να τονίσω κάποια στοιχεία που περιγράφουν την ρυθμιστική μας προσέγγιση και τις βασικές αρχές των ευρωπαϊκών κανονισμών. Η εξασφάλιση της ασφάλειας προφανώς, αλλά ταυτόχρονα η ανάπτυξη της αγοράς είναι ουσιώδης. Η ασφάλεια και των τρίτων μερών στο έδαφος, αλλά βεβαίως η ασφάλεια των επιβατών είναι πρωταρχική. Εμείς στηρίζουμε την επιλογή της ΕΑΣΑ στην τεχνική της νομοδότηση σχετικά με τις τεχνικές επιχειρήσεις. Και βασιζόμαστε σε δύο σενάρια σχετικά με τις τεχνικές αυτές επιχειρήσεις συγκεκριμένα που δίνουν ένα σαφές πλαίσιο στους φορείς και μειώνουν το ρυθμιστικό άχθος για τις ε, αρχές ε, της πολιτικής αεροπορίας. Χρειάζεται ευελιξία, βεβαίως, η αγορά στηρίζεται από την καινοτομία, οι υπηρεσίες εξελίσσονται. Αν ο κανονισμός δεν μπορέσει να παρακολουθήσει το ρυθμό αλλαγών που σημειώνονται στην αγορά, αυτές οι προσαρμογές δεν θα μπορέσουν να είναι επικαιροποιημένες. Χρειάζεται μια προσέγγιση από βάση του κινδύνου και ο κανονισμός δεν μπορεί να επαναλαμβάνει προηγούμενες διατάξεις. Δηλαδή οι διατάξεις σχετιζόμενες ε, με τον τηλεχειρισμό δεν μπορούν να είναι αντίστοιχες με αυτές που ήταν στο παρελθόν. Ε, επίσης χρειάζεται κάποιο είδους επικουρικότητα ώστε να αναπτυχθεί η αγορά σε όλη την Ευρώπη αλλά και να εξεταστούν κάποια τοπικά εμπόδια η κοινωνική αποδοχή των ε, πτήσεων πάνω από ε, κατοικημένες περιοχές όπως και οι στρατιωτικές ε, δραστηριότητες εκπαίδευσης που δεν είναι ίδια ένταση σε κάθε χώρα. δεν μπορούμε να έχουμε ενιαία απάντηση απέναντι στις διάφορες πτυχές των δραστηριοτήτων αλλά χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και ένα κοινό πλαίσιο. Δεν αναφέρθηκα ακόμα συγκεκριμένα σε θέματα ασφαλείας. Οι αυξανόμενες περιπτώσεις drones που έχουν σημειωθεί και ταυτοποιηθεί στο 2015 τονίζουν την ανάγκη συμμόρφωσης σχετικά με τις πτήσεις πάνω από κατοικημένες περιοχές και κυρώσεις. Ο Πρωθυπουργό ανέθεσε μία υπουργική εξέταση και συστάσεις που θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο σχετικά με την ε, χρήση στην πολιτική αεροπορία drones στη Γαλλία. Οι βασικέ τάσει είναι οι εξής. Υποχρέωση για τους παραγωγούς και εισαγωγή σε κάθε τέτοιο αεροσκάφος να επισυνάπτουν τους κανόνες και τις συστάσεις χρηστής συμπεριφορά. όπως επίσης και για την ε, πτήση πάνω από συγκεκριμένε περιοχές. Θα χρειάζεται επίσης μια ηλεκτρονική ταυτότητα κάθε τέτοιου αεροσκάφους και προτάθηκε από την Γαλλική Γερουσία μια σειρά αποστάσεων που συμπεριελάμβαναν και διατάξεις για τεχνικούς περιορισμούς. Σας ευχαριστώ που μας επιτρέψατε να συμμετάσχουμε σήμερα. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Ο Λουκ παρακαλώ, από την ΕΑΣΑ. Έχετε τον λόγο. Um, Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους σας. Αυτό που θα θέλαμε να σας πούμε εδώ είναι ότι φυσικά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη ευθυγραμμίζονται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με τις προτάσεις της ΕΑΣΑ για τον καθορισμό ενός πλαισίου ασφάλειας για τις ενέργειες μεταφόρες. Δεδομένου όμως του γεγονότος της, του επίλυδος αυτής της νέας αφήξεως σε ένα σύνθετο πλαίσιο. Υπάρχει ανάγκη, όπως αναφέρθηκε από προλαλήσαντα, να καθοριστεί με ακρίβεια τι θα ισχύει για τις διαφορετικές κατηγορίες. Χαμηλός κίνδυνος, μέσου επίπεδου κίνδυνος και υψηλού επίπεδου κίνδυνος όσον αφορά την δραστηριοποίηση των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Πρόκληση λοιπόν πρώτα να δούμε πώς μπορεί μια τέτοια προσέγγιση ανακατηγορία να λειτουργήσει και να ισχύσει και θα θέλαμε σε μεγάλο βαθμό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συνολική προσέγγιση ώστε όλοι από πλευράς βιομηχανίας και όσων θα εμπλέκονται στη λειτουργία αυτών των αεροσκαφών να υποχρεούν να λειτουργήσουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Δεύτερο σημείο, αυτό ήταν το πρώτο. Συχνά οι ρυθμιστές όταν αρχίζουν να ρυθμίζουν ε, καταστάσεις έχουν καθυστερήσει ήδη σε σχέση με τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Δεν, αυτό δεν ισχύει μόνο στον τομέα των, ε, της, ε, των αερομεταφορών. Είναι το θέμα της καθυστέρησης ε, του ρυθμιστικού έργου. Το να συνεργαστούμε όλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο λοιπόν είναι η ενδεδειγμένη λύση για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα με τον πιο κατάλληλο τρόπο να υπάρξουν οι αναγκαίοι ορισμοί ώστε να ανταποκριθούμε στα επίπεδα ασφάλειας που απαιτούνται. Λοιπόν, αυτό το οποίο κατά κάποιο τρόπο σίγουρα θα θέλαμε να επιτευχθεί είναι πολύ σημαντικό να εργαστούμε ταχύτατα με ταχύς ρυθμούς, ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε στους ευρωπαϊκούς εθέρες τα μη πανδρομένα αεροσκάφη. Υπάρχουν ε, πολλές προσδοκίες ε, και θα πρέπει να δράσουμε εντάχει, ταχύτατα, πολύ γοργά, για να δημιουργηθούν ε, οι πιο ενδεδειγμένες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτό, για να μπορέσουμε αυτό ανακράτως αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο να δράσουμε, ώστε να υπάρξει ένας κοινός παρονομαστής, να μπορέσουμε να βρεθούμε πολύ κοντά σε αυτά τα οποία ανέφερε ο προλαλής Υπάρχει ανάγκη να δράσουμε από κοινού για να καθορίσουμε τους περιορισμούς που θα πρέπει να ισχύουν ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το πλαίσιο το ασφαλείας, το πλαίσιο ασφαλείας με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Να υπάρχει λοιπόν έλεγχος αποτελεσματικός των κινήσεων αυτών των αεροσκαφών και γι' αυτό θα χρειάζονται προδιαγραφές από πλευράς των βιομηχανιών βιομηχανικές προδιαγραφές ε, εξορισμού αυτό πρέπει να γίνει από τις βιομηχανίες ώστε να υπάρξει μια εκτίμηση, ένας, ε, μια μελέτη και εκτίμηση κινδύνων ε, που θα απορρέουν, ώστε να μπορέσουν να προταθούν μέτρα αντισταθμιστικά για την ασφάλεια. Το ερώτημα το οποίο διατυπώθηκε πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Φυσικά η εφαρμογή είναι κάτι διαφορετικό πρέπει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο και επ' αυτού δεν υπάρχει καμιά ένσταση ή αντίρρηση ώστε να υπάρξει μια συνολική εποπτεία για το πώς θα μπορέσουν αυτά να λειτουργήσουν. Σε τοπικό επίπεδο είναι καλύτερο να υπάρχει αναλογική εφαρμογή σε σχέση με τις ε, προσδοκίες. Εκείνο που απαιτείται είναι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση να καθοριστούν τα μέσα και εργαλεία τα οποία θα διατεθούν από τις ε, βιομηχανίες ώστε να υπάρξουν οι ε, περιορισμοί και οι διατηρήσει διατάξεις που θα διέπουν το πεδίο αυτό. Κάτι το οποίο θα πρέπει, θα πρέπει να βαίνει εκ παραλίλου με την πρώτη προσπάθεια ενώ εν τω μεταξύ είναι εξίσου σημαντικό να υπάρξουν συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας ώστε να, γνωρίζουμε πώς διαμορφώνονται οι κίνδυνοι και να μπορούν ε, να επιβληθούν σε όσους ε, λειτουργούν τέτοια, ε, δρούν με τέτοια αεροσκάφη να επιβάλλουμε τις, τους κανόνες εκείνους που είναι αναγκαίοι. Το βλέπουμε και το, με δημοσιεύματα του τύπου ότι υπάρχουν καθημερινά τέτοια ε, συμβάντα, πολλές φορές ε, που μπορεί να οδηγούν και σε ατυχήματα σε σχέση με ένα ε, σύστημα που απαιτείται για την ασφάλεια. Τέτοιου είδους συμβάντα θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε μια κεντρική αρχή ώστε να γνωρίζουμε το τι συνέβη και να μπορούμε να συναγάγουμε συμπεράσματα για το τι πρέπει να γίνει ευρωπαϊκά σε σχέση με κράτη για παράδειγμα που δεν έχουν την ίδια πείρα και τεχνογνωσία όπως ε, τα υπόλοιπα. Ένα άλλο στοιχείο που θα ήθελα εδώ να αναφέρω είναι η ανάγκη να υπάρξει, να μπορέσει να καταδειχθεί με σαφήνεια ότι τα μη πανδρομένα αεροπλάνα, ε, αεροσκάφη, δεν είναι η μόνη περίπτωση. Όταν για παράδειγμα είχαμε αερόπλια ή αερόστατα ε, που σε, πρέπει οι κανονισμοί να εναρμονίζονται πρέπει να βλέπουμε πώς είναι δυνατόν να, σε ένα ενιαίο πλαίσιο να υπάρχουν κανονισμοί και από τέτοιου είδους παραδείγματα να εμπνευστούμε και να πορευθούμε για την ρύθμιση αυτού του τομέα των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Και μια τελευταία παρατήρηση, σίγουρα πολύ σημαντική και αυτή επίσης είναι ότι όταν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη αρχίσουν να λειτουργούν στους ευρωπαϊκούς εθέρες σημαντικό είναι για όσους εμπλέκονται ή για τις ε, βιομηχανίες ε, να μην ε, υπάρχουν μόνο εθνικές διατάξεις και κανονισμοί που θα συνεπάγονται και υψηλό κόστος ε, σε σχέση με τις βιομηχανίες ε, και να δούμε και πώς εδώ θα μπορούν ε, οι βιομηχανίες να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο θετικό και γι' αυτό σε σχέση με τους όσους εμπλέκονται για τους ορισμούς που θα πρέπει να καθοριστούν θα πρέπει από κοινού με τις βιομηχανίες να δράσουμε ώστε να ρυθμίσουμε αυτό το τομέα όπως απαιτείται. Πρόεδρος σας ευχαριστώ και πάλι σας ευχαριστούμε και τους τέσσερις ε, που ε, μας εκθέσατε τις απόψεις σας. Θέλω και μια ομάδα επισκεπτών να καλωσορίσω από την ε, Ομοσπονδία, Εθνική Ομοσπονδία de, Transport, de, που βρίσκονται εδώ στην Επιτροπή μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ. Jetzt hat Τώρα, Γκαμπριέλε Πρόεδρε, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ίδιο τον εισηγητή, λέει η κυρία Πρόης από την ίδια πείρα των προηγούμενων εβδομάδων γνωρίζω πόσο σύνθετο και περίπλοκο είναι το θέμα αυτής της έκθεσης και είναι θετικό το ότι υπάρχει μια τέτοια καλή συνεργασία. Υπό το πρίσμα των σοσιαλδημοκρατών θέλω να θέσω μια ανάποψη εδώ στο προσκήνιο. Δηλαδή σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρέπει εδώ να καλύψει ένα κενό. Έχουμε πολλές επιδεινωμένες προϋποθέσεις όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα στις εναέριες μεταφορές. Γι' αυτό οι τροπολογίες μας αφορούν τη διασφάλιση ενός θετικού πλαισίου στις αερομεταφορές σε διάφορα σημεία. Προτείνουμε μεταξύ άλλων ένα νέο άρθρο ώστε να ε, ε, εξετάζεται αυτό το θέμα ξεχωριστά και να ρυθμίζεται ξεχωριστά. Όσον αφορά την έκθεση γενικά, εκθέτω την άποψη ότι η ΕΑΣΑ θα πρέπει να ενισχυθεί, να ενδυναμωθεί στις αρμοδιότητές της, ώστε να επιτευχθεί πρόσθετη αξία ε, στην ασφάλεια ώστε ε, θα πρέπει από την άλλη πλευρά να αποφύγουμε ε, διπλοεπικάλυψη ε, όσον αφορά διάφορες διατάξεις. Για το άρθρο 76 συμβουλευτικές δραστηριότητες όσον αφορά θέματα ασφάλειας ή όσον αφορά σύναφη θέματα. Ανεξάρτητα από αυτό η αξιολόγηση κινδύνων κατά πρώτο λόγο πρέπει να διασφαλίζεται από τα κράτη-μέλη. Εδώ θα πρέπει σε σχέση με τον εξοπλισμό και με τα δίκτυα να δράσουν ώστε να δημιουργηθεί αυτό το πλαίσιο. Το ίδιο και για το περιβάλλον. Θα πρέπει οι διασυνδέσεις σε σχέση με το περιβάλλον να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης και να αναφερόμαστε σε διεθνείς προδιαγραφές που έχουν ήδη συμφωνηθεί σχετικά. Αυτό αφορά και την εντολή της ΕΑΣΑ που θα πρέπει να καθορίζεται με απόλυτη σαφήνεια. Όμως είμαστε υπέρ της διασφάλισης της ποιότητας μέσω της εντολής της ΕΑΣΑ και για την κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων ώστε να μπορέσουν να υπαρκέσουν οι δεξιότητες και οι ικανότητες τους. Performance-based regulation, δηλαδή ρυθμίσεις που θα στοχεύουν στην λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα ώστε η ασφάλεια στο μέλλον να έχει προτεραιότητα. Γι' αυτό είμαστε υπέρ μιας ρύθμισης που θα είναι αναλογική και συνετή, ώστε να είναι λειτουργικά τα όσα θα προτείνουμε και να μπορέσουμε τις αναγκαιότητες, τις ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν με αποτελεσματικό τρόπο να τις ρυθμίσουμε η ευρωπαϊκή ε, προσέγγιση σε σχέση με την προσέγγιση των κρατών μελών για να υπάρχει εδώ η δυνατότητα αυτή πρέπει εθελοντικού χαρακτήρα να είναι αυτή η συμφωνία ώστε μέσω ε, συνεργασίας αυτής της αρχής και των κρατών μελών να υπάρξει η καλύτερη αποτελεσματικότητα. Τίθεται τώρα εδώ το ερώτημα ποιο δυναμικό θα έχει η ΑΣΑ; Θέλω να τονίσω από αυτή τη θέση ότι μια και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, ταχύτατες εξελίξεις στις ε, τεχνολογικές, ε, ε, στα τεχνολογικά επιτεύγματα δεν πρέπει να υπάρξουν περικοπές κονδυλίων. Είναι αναγκαία με βάση το αντίστοιχο άρθρο, με βάση τις προτάσεις για τα κονδύλια αυτά να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τα αναγκαία μέτρα. Παραμένουν όμως και κάποια ερωτηματικά. Πώς θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα μελλοντικά έργα και καθήκοντα για τα τέλη τα οποία θα πρέπει να εισπράττονται, για παράδειγμα αυτό το Eurocontrol, για να μπορέσουν να, να υλοποιηθούν όλες αυτές οι υποχρεώσεις μας. Σημαντικό είναι οι μικρότεροι εμπλεκόμενοι σε αυτόν τον τομέα να μην αφαιθούν εκτός πλαισίου και έχουμε και αντίστοιχε τροπολογίε προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι ε, χάρη να αναψυχή ασχολούνται με τι ε, ε, ε, με μικρά αεροπλάνα και αυτοί πρέπει να καλύπτονται. Πρέπει να εργαστούμε νομοθετικά εκεί όπου υπάρχει ανάγκη να ρυθμίσουμε πράγματα. Με τον κανονισμό εδώ λοιπόν πρέπει να λάβουμε υπόψη και το άρθρο 123 συγκεκριμένα. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ρυθμίσεις ε, σε σχέση με ε, προηγούμενες, ε, ε, προηγούμενους κανονισμούς θα πρέπει να υπάρξει μια διευκόλυνση και ελάφρυνση του έργου. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε ότι μια και αυτό δεν ανήκει σε αυτό το πλαίσιο με τον καλύτερο τρόπο θα πρέπει να διαγραφεί. Έχουμε σημαντικές προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουμε για αυτό το χατοφυλάκιο τις επόμενες εβδομάδες. Προσδοκώ να δω ποια θα είναι η τελική έκβαση με τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο ασφάλειας για τις μελλοντικέ μας δράσεις σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε πολύ τους επαΐοντες για τα όσα μας εξέθεσαν για τα μη επανδρομένα αεροπλάνα που είναι ένας άγνωστος σχετικά τομέας και οι προτάσεις τους είναι πολύ θετικές. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ για όσα μας εκθέσατε. Τζάκη <clears throat> Κώστα παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Και να έλθω στα μη επανδρομένα, στα drones και στις τελευταίες ε, μου παρατηρήσεις θα αναφέρω αυτά που θέλω να πω για αυτό το θέμα. Προποποιεί ο κ. Μαρινέσκο την έκθεση κομισιών. Θέλω λοιπόν πρώτα να σχολιάσω κάποια σημεία αυτή τη πρόταση και μετά να έλθω στα μία επανδρομένα. Είναι προφανές ότι ορισμένες από τις τροπολογίες ε, του εισηγητή ε, θα τις στηρίξουμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες που για συγκεκριμένους λόγους μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να τις στηρίξουμε. Υπάρχει μια αναφορά σε όλη την έκθεση ε, που αλλάζει την έμφαση ε, από την αρμόδια αρχή στον οργανισμό. Σε 61 τροπολογίες περίπου. Και αυτό δεν μπορούμε να το στηρίξουμε, διότι δεν είναι δική μας δουλειά εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουμε μικρομάνατζμεντ, μικροδιαχείριση του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί ο κανονισμός αυτός, ε, οι αρχές ε, της, ε, των αεροπορικών μεταφορών, η ΔΟΠΑ, ο Διεθνής, η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας. Δεν είναι δική μας δουλειά. Εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πάρουν πολύ σοβαρά υπόψη τις ευθύνες και οι λεπτομέρειες είναι δική τους δουλειά καθαρά. Ε, άρα ε, δεν θέλουμε να αλλάξει καθόλου αυτή η ορολογία από competent authority να μιλάμε για agency. Τώρα, ε, ο οργανισμός έχουμε τα θέματα του καταστατικού, αν αλλάξει ονομασία. μπορεί να έχουν ε, υπάρξει κάποιες εθνικές διατάξεις υπό το ακρονίμιο ΕΑΣΑ. Και ο οργανισμός έχει αυτό το όνομα σε διεθνές επίπεδο. Το να αλλάξουμε το όνομά του λοιπόν και να το λέμε European Aviation Agency δεν είναι κάτι καλό. Έχουμε την ΕΜΖΑ για την θαλάσσια ασφάλεια, την ασφάλεια στην αεροπορία και έχουμε και την ΕΑΣΑ. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η λέξη safety μέσα. Γιατί είναι στο επίκεντρο ε, του έργου αυτού του οργανισμού. Αυτά τα δύο λοιπόν που είναι πιο πολύ γλωσσικής ε, φύσεως σχόλια. Να συμφωνήσω τώρα με την τροπολογία 14 του κυρίου Μαρινέσκου για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Φυσικά θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου ο οργανισμός ή οποιοδήποτε άλλος ε, μπορεί να προτείνει μια κατεξουσιοδότηση πράξη, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να είναι ένα τετελεσμένο γεγονός για όλους τους τομείς που καλύπτουν σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επιλαμβάνονται τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδεχομένω και να συζητούμε εδώ κάποια πράγματα που άπτονται τη εφαρμογή. Ε, να μιλάμε για πιο πολυεκτελιστική πράξη, ίσω και όχι κάτι εξουσιοδότηση. Τώρα, στο σχέδιο της Κομισιόν, δεν υπάρχει πλέον καμία αναφορά ε, στον ΙΚΑ όταν μιλάμε για τις εκπομπές και το θόρυβο. Θα θέλαμε να έχουμε τις αναφορές ε, στον ΙΚΑΟ. Όχι μόνο στην αρχή, αλλά σε όλο το έγγραφο, εκεί που πρέπει, για τα πρότυπα που ισχύουν. Αυτό πρέπει να ισχύει, διεθνή πρότυπα. Αλλιώς δεν θα υπάρξει καμία ε, βεβαιότητα στον κλάδο. Για το εκτελεστικό, ε, το executive board, δεν το χρειαζόμαστε. Management board αρκεί. Γιατί να προσθέσουμε ένα ακόμα στρώμα γραφειοκρατίας. Δεν θα υπάρξει κάποιο κέρδος για κανέναν. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, το άνοιγμα διεθνών γραφείων. Καλή ιδέα, πολύ καλή. Όχι παντού βέβαια, διότι φυσικά υπάρχει εκπροσώπηση στην ε, Ουάσιγκτον και στον Καναδά, στην ΔΟΠΑ υπάρχει. Ίσως Συγκαπούρη, Ντουμπάι και σημαντικές περιοχές που είναι καλό να υπάρχει εκπρόσωπος εκεί. Σε ό,τι αφορά τώρα την χρηματοδότηση, υπάρχουν κάποια τέλη ε, που τώρα τα παίρνει το Eurocontrol. Το να πάνε στον οργανισμό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Όπως γνωρίζετε, εγώ στηρίζω την ε, χρηματοδότηση του ΕΑΣ για να ξέρει πού κινείται με τον ε, προπολισμό. και θέλω μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση γιατί το 25% προέρχεται από τον κλάδο. Είμαι υπέρ λοιπόν, αλλά δεν νομίζω ότι μια απάντηση αυτό προτείνεται εδώ. Δεν ξέρω ποιος το προτείνει βέβαια. Τώρα, στα θέματα της ασφάλειας είναι πολύ ακαθόδηστο ζήτημα. Ε, σε σχέση με την αεροπορία. Πώς θα μπορούσε να διατυπωθεί στην αναθεώρηση αυτού του κανονισμού. Μήπως ήταν καλύτερη εθελοντική συνεργασία δεδομένων των δυσχεριών και των τρομοκρατικών επιθέσεων για κάποιον άλλον συμβάντων της περσινής χρονιάς. Το θέμα είναι πώς θα διατυπωθούν όλα αυτά. Καταλαβαίνω το στόχο. Εν τέλει, όσο αφορά την εποπτεία, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σωστή εποπτεία. Αλλά οι επιχειρήσεις, οι εταιρείε που ζητούν θα πρέπει να ορίσουν και ποιο θα είναι αυτός που θα αναλάβει την εποπτεία το κράτος μέλος ή ο ΕΑΣΑ. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ομαλή ε, λειτουργία εδώ ε, και να μην υπάρχουν άλλοι επικαλύψεις. Αυτά για τον εισηγητή και έρχομαι στα drones. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι πάνω από ένα χρόνο εργαστήκαμε πάνω στην έκθεση για τα μη επανδρομένα. Υπάρχει αυτή η έκθεση. Είχα πάρα πολύ ε, διεξοδικές συζητήσεις ε, και με τον πρόεδρο του Τζάρ, τον κλάδο, ε, τους ελεγκτές, ε, το τμήμα των μεταφορών, φυσικά με τον έαζαμε την Ένωση των ε, ε, Κυβερνητών Αεροσκαφών, μιλήσαμε με άτομα από την Ουάσιγκτο κτλ. κτλ. Άρα υπήρχε ένα πολυερέστατο feedback γιατί θέλαμε να ξεκινάμε όλα από την ίδια βάση και νομίζω ότι η έκθεση ήταν πάρα πολύ καλή, εξαιρετική. Όλα τα σημεία που έθεσαν λοιπόν οι προσκεκλημένοι μας και χαίρομαι να, που βλέπω που βρισκόμαστε τώρα έξι μήνες μετά, όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα. Όλα όσα είπατε όμως εμείς στην Επιτροπή μας τα έχουμε θέσει ήδη επιτάπητος ε, για την αεροπλοημότητα, την πιστοποίηση, εμπορική χρήση, χρήση αναψυχής, ε, την ταυτοποίηση, τον κάτοχο, την καταχώρηση, ε, ε, την κατεκπαίδευση, όλα αυτά που είπατε, geofencing, no-flight zone, επίπεδα κινδύνου, χαμηλό έψαλο κτλ. κτλ, κτλ. Και φαντάζομαι θα υποστηρίξει και ο πρόεδρος, γιατί είχαμε πληρέστατες συζητήσεις που έγκυται ανησυχία μου όμως σχεδόν 700 ευρωβουλευτέ υποστήριξαν αυτή την έκθεση και έδειξαν την κατεύθυνση που θέλουμε εσείς οι ρυθμιστές να ακολουθήσετε. Φυσικά η προσέγγιση βασίζεται στον κίνδυνο. Φυσικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη διεθνής διάσταση. Δεν μιλάμε για δύο συνοριακό επίπεδο. Πρέπει και οι κατασκευαστές να βρουν όλη αυτή την ε, ε, κατάλληλη τεχνολογία, τα τσί, το geofencing Είναι ε, αυτό που μας ενδιαφέρει ε, όμως το κεντρικό κομμάτι και όχι η κορυφή. Είμαι μεν αισιόδοξη, όμως ε, δεν μπορώ να γκρύψω την ενόχλησή μου από αυτά που άκουσα σήμερα. Έξι μήνες μετά μιλάει κανείς με κανέναν άλλον. Έχουμε καλούς εκπροσώπους από διαφορετικούς οργανισμούς, φορείς. Όλοι έχουν λάβει μέρος σε αυτή τη συζήτηση για τα drones. Άρα φαίνεται να μην μπορείτε να κάνετε κάτι. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι πάντα υπάρχει λύση. Πάντα μπορεί κάτι να γίνει. Άρα όταν έρθει κανείς την επόμενη φορά να μας ενημερώσει, καλό θα ήταν να μας μιλήσει και για το πώς ε, και τι γίνεται συγκεκριμένα. Το θέμα είναι πολύπλοκο και αυτό το κατανοούμε. Όμως ε, ε, η εθνική επιβολή της νομοθεσίας είναι σημαντικό θέμα. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε αυτούς που δημιουργούν προβλήματα με τη χρήση ε, drones, με τη λειτουργία drones. Εμείς λοιπόν αναζητούμε λύσεις πάντα και κάποια στιγμή θα ήθελα να ακούσω και από εσά λύσεις. Και εδώ θα ολοκληρώσω ε, κύριε Πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι ήταν σημαντικό ε, όλοι οι προσκεκλημένοι που έρχονται εδώ, επειδή ξέρουν ότι αυτό το θέμα είναι στην διάταξη, να έχουν αντιληφθεί ότι εδώ και πολλούς μήνες, 18 σχεδόν, πάνω από χρόνο λοιπόν, ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Είπε και ο κύριος Μαρινέσκο ότι θα ξανασυναντηθούμε οι σκιώδεις ηγητές σε μια προσεχή συνεδρία και ελπίζω να έχουμε μια έκθεση η οποία ε, θα επιτύχει τους στόχους της και θα μπορέσει να βοηθήσει ε, να έχουμε ένα αποτελεσματικό οργανισμό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Μίτενμπεκ παρακαλώ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινέσκο για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεση ε, που εξεπώνησε. Είναι σίγουρα δύσκολη δουλειά να αξιολογηθούν όλα τα τεχνολογικά στοιχεία, αλλά είναι και πολύ μεγάλη σπουδαιότητα, διότι η ασφάλεια είναι ιδιαίτερα σπουδαίο ζήτημα όταν έχουμε τα θέματα των ε, μεταφορών λειτουργική και αποτελεσματική άσα είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών και σε σχέση με την ευρωπαϊκή βιομηχανία αερομεταφορών. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις δικές μας χωριστές προδιαγραφές ε, που θα ακολουθούν ε, την οργάνωση ΑΙΚΑΟ στο Μοντρεάλ, αλλά όχι αποκλειστικά μόνο αυτό. Πρέπει να είμαστε και εμείς ε, να εμπνευστούμε και να δημιουργήσουμε τέτοιες προδιαγραφές. Ασφάλεια. Ασφάλεια με κεφαλαία είναι τεράστια σημασία ε. Και για το άρθρο 76, για παράδειγμα, τον κανόνα 76, όπου η ΆΣΑ θα μπορεί να έχει αρμοδιότητα για την κυβερνοασφάλεια και η ιδέα να ρυθμιστούν ε, οι ζώνες ε, σειράξεων. Ε. Να αναλάβουμε λοιπόν την αναγκαία πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Απαιτείται συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΑΣΑ. Μεγάλη σπουδαιότητα και εμβέλεια σε αυτό για να διασφαλιστούν τα θέματα ασφάλειας. Βλέποντας τις τροπολογίες έχουμε μια θα έλεγα εξαιρετική, πολύ καλή προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων ενισχύοντας τον διεθνή ρόλο της ΕΑΣΑ σε σχέση με τρίτες χώρες και τον ενεργό ρόλο της ΕΑΣΑ όταν θα έχουμε θέματα ελέγχου εναέριων μεταφορών. Πρέπει να δούμε στην εφαρμογή φυσικά όλα αυτά εξειδικευμένα, αλλά η ιδέα είναι πολύ καλή. Είμαι λιγότερο ικανοποιημένος με τις άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν από τον κύριο Μαρινέσκου σε σχέση με το άρθρο 1 για παράδειγμα. Και εδώ πρέπει να πω ότι η ασφάλεια, οι υψηλά επίπεδα ασφάλειας πρέπει να βαίνουν εκ παραλίλου με τα θέματα περιβαλλοντικής ασφάλειας. Η διαπίστευση επίσης ε, ε, των εθνικών συλλόγων οργάνων για την ασφάλεια ε, μεταφορών πρέπει να μην υπερβούμε τα εύθετα πλαίσια και υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να επεκταθούμε περισσότερο και να τα δούμε πιο εξειδικευμένα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές τροπολογίες ε, που ε, μέσα στο πλαίσιο της προσπάθειας να υποστηρίξουμε ε, τις σωστές κατευθύνσεις δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε. Εδώ ο προϋπολογισμός ε, και τα καθήκοντα της ε, ΕΑΣΑ είναι σημαντικότατα θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν και θα καταθέσουμε τροπολογίες και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν έχουμε τα θέματα των ε, καθηκόντων και τα κονδύλια από πλευρά Πρέπει να δούμε ότι υπάρχει η επέκταση του ρόλου σε άσα είναι ένα πολύ καλό βήμα προς τα εμπρός, όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι σε θέση με βάση τα κονδύλια που θα διατεθούν να αντιμετωπίσει τα καθήκοντά της η θα πρέπει να συνεχίσουμε να συσσωρεύουμε και να προσθέτουμε όλο και περισσότερες αρμοδιότητες και καθήκοντα στην ΕΑΣΑ χωρίς να υπάρχουν τα αναγκαία κονδύλια που θα συνοδεύουν ε, όλα αυτά τα θέματα. Επίσης και το θέμα της, ε, των ε, υπηρεσιών, επίγειων υπηρεσιών. Είναι πολλά θέματα στα οποία πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Δεν επεκτείνεται ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επέκταση αρμοδιοτήτων πρέπει να τεκμηριώνεται με τον καλύτερο τρόπο και χρηματοοικονομικά από πλευράς Eurocontrol και EASA πρέπει να καθοριστούν και να αποσαφινιστούν πολλά θέματα. Και για την μελέτη επιπτώσεων για παράδειγμα και όσον αφορά την χρήση των τελών διαδρομών για να ε, χρηματοδοτηθούν οι δραστηριότητε τη ΕΑΣΑ δεν υπάρχουν όμως αντίστοιχες ε, πτυχές που να καθορίζουν αυτές τις συνιστώσεις από πλευρά της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο καθορισμός από πλευράς βιομηχανιών ε, του θέματος τέτοιων τελών ίσως θα μπορούσε να είναι χρήσιμος. Πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρξουν δίπλο επικαλύψεις μεταξύ ΙΑΣΑ και Eurocontrol όσον αφορά τα καθήκοντά τους και να μην πληγεί διτά, να μην πληγούν οι βιομηχανίες διτά λόγω τέτοιων τελών. Τώρα για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι το Ευρωκοινοβούλιο έχει πολλές πρωτοβουλίες ε, που ε, έχει αποδηθεί, απεκδηθεί και έχει αναλάβει. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει η ασφαλής ένταξη στην αεροβιομηχανία των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Χρειάζονται κανόνες και κανονισμοί για αυτά τα αεροσκάφη. Χρειάζεται επίσης αξιολόγηση κινδύνων, να δούμε την εφικτότητα και το, ε, τις δυνατότητες που έχουμε να χρησιμοποιηθούν τεχνολογικά τέτοιου είδους δυνατότητες. Πρέπει να διασφαλιστούν ε, ότι οι περιορισμοί που θα υφίστανται σε σχέση με τον ε, ε, αεροχώρο, με τους εθέρες και τα αεροδρόμια πρέπει να ισχύουν ώστε να αποφευθούν συγκρούσεις ε, στους εθέρες. Ε, χρειαζόμαστε προτάσεις ε, ώστε τα σημεία εκείνα που πρέπει να ρυθμιστούν να μπορέσουν να διευθετηθούν, να μπορέσουμε να ε, συμπτύξουμε και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με τις προτάσεις που θα καταθέσουμε. Πρέπει να υπάρξει ασφαλής ένταξη των μη επανδρομένων αεροσκαφών στην ευρωπαϊκή αεροναυπηγική και βιομηχανία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έχετε τον λόγο τώρα εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον ε, κύριο Μαρινέσκου για την ε, γνωμοδότησή του. Πολλές από τις τροπολογίες μπορούμε να τις, εγώ θα μπορούσα να τις υποστηρίξω και θα ήθελα να σημειώσω κάποιες λεπτομέρειες αυτό που είναι πιο ανησυχητικό θεωρώ ότι είναι η πρόταση αλλαγής του ονόματος οργανισμού. Διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια δόκιμη επιχειρηματολογία σχετικά με την πρόταση αυτή που θα οδηγήσει σε αυξανόμενο κόστος γιατί πρόκειται για έναν αναγνωρισμένο διεθνώς οργανισμό ε, και το σύνολο των νομοθετημάτων και διατάξεων ε, ε, αναφέρονται παραπέμπουν στο όνομά του. Δηλαδή μας φαίνεται κάπως τραβηγμένο να αλλάξουμε το όνομα του κανονισμού έτσι απλώς για να το αλλάξουμε. Χρειάζεται πολύ περισσότερη οικονομική ανάλυση. Επίσης δεν θα ήθελα να αφήσουμε τις περιβαλλοντικές πτυχές εκτός του κειμένου, όπως κάποιες τροπολογίες προτείνουν. Δηλαδή να παρακάμψουμε όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, δεν είναι πολύ καλή ιδέα αυτή και να ρωτήσω και το εξής για το άρθρο 72. Τι, ποια είναι η πρόθεση αυτής της ε, τροπολογίας. Γιατί δεν αντιλαμβάνομαι αυτό το σύστημα προστήμων ή κυρώσεων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. αυτό θα μπορούσε να φτάσει και στο επίπεδο του προσωπικού των υπαλλήλων ή μόνο της διοίκησης. Και επίσης ποια είναι η επιχειρηματολογία πίσω από την ε, πρόταση αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάντως όλους τους εμπειρογνώμονες για τα μία παδρομένα, τα drones και ελπίζω όλοι οι παριστάμενοι, όλοι οι συνάδελφοι στην αίθουσα να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα ζητήματα αυτά, όχι μόνο υπό την έννοια της ασφάλειας, αλλά και υπό την έννοια της ενίσχυσης του συνολικά του τομέα και της εμπειρογνωμοσύνης εδώ. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι υπό τους οποίους θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα μία επανδρομένα αυτά σκάφη με διάφορους τρόπους και πραγματικά ε, τα πρώτα βήματα πραγματοποιούμε εδώ. Όμως ο κανονισμός, η πρόταση κανονισμού έχει ήδη μείνει πίσω. Θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ καλύτερα υπόψη ε, στην ε, νομοθετική μας δουλειά συνολικά όλες αυτές οι εξελίξεις της τεχνολογίας. και θα ήλπιζα ότι θα μπορούσε να διεξαχθεί ένας ε, διαρθρωμένος διάλογος μεταξύ εμπειρογνωμόνων ώστε να μην πλήττεται η ασφάλεια αλλά ανοίγοντας και την δυνατότητα για περαιτέρω καινοτομία εδώ. Ευχαριστούμε. Εσείς έχετε τώρα τον λόγο παρακαλώ. Euh, euh, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η γνωμοδότηση είναι πολύ πυκνή θα προσπαθήσω από όλα αυτά τα στοιχεία να συνοψίσω τα πιο σημαντικά. Ένα στοιχείο ικανοποίησης υπό την οικολογική τουλάχιστον πτυχή είναι η διασύνδεση που τονίζεται μεταξύ της ασφάλειας και του περιβάλλοντος. Αυτή η υπογράμμιση. Το περιβάλλον είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει συνολικά ο κλάδος θα πρέπει να προσαρμοστεί ο κλάδος σε όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν συμβεί την τελευταία περίοδο. Και επίσης έχουμε και μια ιστορική εξέλιξη, θα έλεγα, που είναι η COP21. Ως προς αυτό λοιπόν θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε τους στόχους ε, μείωσης εκπομπών και απομάκρυνση από τον άνθρακα, αλλά είναι σαφές ότι δεν θα είναι η ικανοποιητική η επίτευξη των στόχων της COP21. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε πιο πέρα. Έχει σημειωθεί μεγάλη εξέλιξη, πρόοδος σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα αεροσκάφη ώστε να είναι πιο ελαφρά. Αλλά μερικά από αυτά τα στοιχεία, το είπαν και οι συνάδελφοι, είναι, δεν είναι προς όφελος της ασφάλειας. Θα χρειαστεί λοιπόν μια πλήρη πιστοποίηση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ναι, αλλά δεν θα υπάρξει διατάραξη της ε, καλής ισορροπίας μεταξύ των ε, πτυχών ασφαλείας και των πτυχών που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την προστασία του. Ένα δεύτερο στοιχείο που έχει σημασία, κύριε Σίγητα, μετά την ασφάλεια και το περιβάλλον, είναι ο σχετισμός μεταξύ των θεμάτων ασφαλείας και αυτή τη φορά των κοινωνικών ζητημάτων. Ο κύριος ε, Πατρίκ Κιάη, ε, τα στοιχεία της πτώσης ε, του ουκρανικού, μάλλον του αεροσκάφους της θύσης στην Ουκρανία, όπως και της αντίστοιχης πτώσης του αεροσκάφους των German Wings, ε, αναφέρομαι σε αυτά γιατί είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Επί τη βάση δηλαδή την πίεση που ασκείται για τις συμβάσεις, για το χρόνο, για την πίεση που αισθάνονται οι πιλότοι, το προσωπικό αεροσκάφους. Υπάρχει ένας αριθμός από στοιχεία, επί τη βάση των οποίων τα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία και η επισφάλεια της εργασίας έχει επιπτώσεις και έχουμε χάσει και αεροσκάφη για τους λόγους αυτούς. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όπως έλεγα, αλλά θα περιοριστώ στην ε, σημερινή ακροασία. Εγώ άκουσα προσεκτικά τόσα είπατε. Θεωρώ ότι το θέμα των drones, των μη επανδρομένων, είναι επίγον. Πρέπει να το δούμε έκτακτα. Πρέπει να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό της χρησιμοποίησής τους και γιατί. Γιατί το, τροποποιούμε τον κανονισμό του ΕΑΣΑ και σε 10 χρόνια, σε 10 χρόνια, 2016 λέει ο κανονισμός από τότε που το λέει, θα είναι μέρος της ζωής μας τα μη επανδρομένα. Τα βλέπουμε να περνάνε πάνω από τους ε, δρόμους, πάνω από τα χωράφια κτλ. Τώρα, καλό είναι να μην το βλέπει κανείς ε, ως ε, απόλυτη απειλή όλο αυτό, έχει και πτυχές ελκυστικές και πολύ ενδιαφέρουσες. Άρα ως το 2026 θα πρέπει να προλάβουμε ορισμένες εξελίξεις. Να έχουμε ένα ελάχιστο πλαίσιο του νομοθετήματος ώστε να ρυθμίζεται η χρήση αυτών των ε, αεροσκαφών. Και λησμονώ το όνομά σας ο κύριος που εκπροσωπούσε τη Γαλλία, την Ντεζέασε, έχετε κάνει πολλές δουλειές και μελέτες επ' αυτού. Αν είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, λάβει κάποιες πρόνοιες σε σχέση και σε συνεργασία και με τα κράτη-μέλη θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπω εδώ έναν ορισμό που λέει ότι drone είναι αεροσκάφος το οποίο εν πάση περιπτώσει τηλεπιλωτάρεται. Πάντως πιλωτάρεται. Οδηγείται από κάποιον. Επομένως θα πρέπει το σύστημα ελέγχου να μπορεί να είναι σε επαφή σε κάθε σχέση με τον άνθρωπο που χειρίζεται και αυτός ο άνθρωπος, ο χειριστής, ο πιλότος, εξ θα πρέπει να έχει την κατάλληλη πιστοποίηση και άδεια. Από την άλλη δεν είναι ακριβώς αεροσκάφος, το drone, με την έννοια του αεροπλάνου. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, αλλά υπάρχουν κοινά στοιχεία με τα κανονικά αεροσκάφη. Υπάρχουν και διαφορές, όπως το πολύ χαμηλό ύψος πτήσης. Υπάρχει λοιπόν διπλός κίνδυνος. Από τα 150 μέτρα οριζόντιος κίνδυνος από τα άλλα αεροσκάφη και σε πιο χαμηλά ύψη εμπόδια του εδάφους. Άρα όλα αυτά τα 0-150 οι κίνδυνοι δηλαδή κοντά στο έδαφος είναι στοιχεία που πρέπει να τα εφεύρουμε γιατί δεν υπάρχουν στις υπόλοιπες διατάξεις για την αεροπορία. Πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν τεχνολογίες ε, αποφυγής εμποδίων να έχουμε μια τράπεζα δεδομένων στην οποία μπορούμε να προστρέξουμε σε περίπτωση προβλήματος ή κινδύνου. Δηλαδή είναι ένα ολόκληρο πεδίο που πρέπει να διερευνήσουμε και πρέπει να βρούμε απαντήσεις σχετικά γρήγορα. Εάν είναι να θεωρήσουμε τα drone όπως αεροσκάφη, ως αεροπλάνα, θα πρέπει να δούμε τις κατηγορίες των μη επανδρομένων εκείνων που παρουσιάζουν τον μικρότερο κίνδυνο και τα οποία θα μπορούσαν ίσως, λέω, ίσως, να χαίρουν κάποιον παρεκκλήσεων, εξαιρέσεων. Θα μπορούσαμε να έχουμε κανόνες για το συνολικό μέγεθος, τον όγκο, τη δυνατότητα ελιγμών του, την ε, επαγγελματική χρήση ή από τη χρήση εκ μέρου ποιου φορέα κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα κανόνα και καμία διαίρεση μεταξύ ομαδοποίηση μεταξύ των ειδών των ντρόουν. Και δεν είναι λεπτομέρεια, το ξαναλέω. Δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της μελλοντική εικόνας των πραγμάτων. Επομένως, σε σχέση με την Επιτροπή θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα όσο γίνεται πληρέστερα. Ο κύριος Μαρινέσκου έχει ήδη πολύ καλά στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πολύ καλή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Μαρινέσκου, σας ευχαριστούμε και εσάς για το έργο σας. Μία ερώτηση παραμένει αναπάντητη για τη διεύρυνση της ε, άσασης αρμοδιότητες της θα υπάρξουν διαφορές μεταξύ των μεγάλων αεροδρομίων που θα είναι διεθνή και των περιφερειακών μικρών αεροδρομίων. Όλα με τον ίδιο τρόπο θα υποστούν αυτές τις επιπτώσεις ή πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση απέναντί τους. Παρακαλώ εσείς έχετε τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ και εγώ από πλευράς μου προς τον κύριο εισηγητή λέει ο κύριος Ερτούγ και από πλευρά των παρεμβάσεων είναι σαφές ότι η σοσιαλδημοκρατική ομάδα υπέρ της καινοτομίας και της ε, λειτουργικότητας από οικονομικής πλευράς ε, τονίζει τις προτεραιότητες. Άσχετα πώς θα δράσουμε πρέπει να πετύχουμε ότι η ΆΣΑ θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία για του ε, τους εθέρες στις αερομεταφορές και να αποφευθούν οι περιττές διπλές υποδομές και διπλοεπικαλύψεις. Ταυτόχρονα πρέπει όμως ε, να διασφαλίσουμε τα νέα καθήκοντα της ΕΑΣΑ με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι λειτουργική. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι στον τομέα της κυβερνοασφάλειας τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει συμβουλευτικός ρόλος από πλευράς της ΕΑΣΑ. Μια και υπάρχει άμεση επίπτωση στην ασφάλεια των, α, της και εδώ θα πρέπει με σαφήνεια τα θέματα των μη επανδρομένων αεροσκαφών να ενταχθούν σε αυτές τις αρμοδιότητες. Ευρωπαϊκά πρέπει να δράσουμε και όχι εθνικά και εμβαλωματικά. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξουν ρυθμίσει και στο εθνικό επίπεδο να εφαρμοστούν. Και αν θυμηθούμε τις άλλες συζητήσεις που είχαμε για διασυνοριακά θέματα, έτσι και στον τομέα της ε, αεροπλοείας, ε, των αερομεταφορών πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ρυθμιστούν τα θέματα των μη πανδρομένων αεροσκαφών. Θα λέγα ότι και εδώ με την ε, παρέμβαση ε, από πλευρά συναδέλφου Πρόης με βάση τις επιδόσεις ε, και την αποτελεσματικότητα πρέπει να προχωρήσουμε. Σε ένα τόσο σημαντικό τομέα όπως στις αερομεταφορές δεν μπορεί η ασφάλεια να υποστεί περικοπές, να συρρυκνωθεί λόγω θεμάτων κονδυλίων ή χρηματοοικονομικών θεμάτων. Εκείνο το οποίο λείπει και απουσιάζει και αναφέρθηκε προηγούμενα είναι ότι εμείς από πλευρά σοσιαλδημοκρατών θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε τους όρους εργασίας των εργαζομένων, επιμόρφωση, κατάρτιση των εργαζομένων που έχουν αρμοδιότητες σε σχέση με τα ίδια τα σκάφη, τα αεροσκάφη. Πρέπει να βελτιωθούν οι όροι απασχόλησης. Δεν είναι λοιπόν αποδεκτό να μην υποβάλλονται προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα και να γίνεται η προσπάθεια με το άρθρο 123 ταυτόχρονα νομοθετικές ε, ρυθμίσεις ε, να εντάσσονται εδώ παρακάμπτοντας, ας το πω έτσι, παρακάμπτοντα, παρακάμπτοντας ε, τις ευθύνες που πρέπει να υπομισθούμε. Εμείς ως σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες πάντα ασκήσαμε επικρίσεις σε τέτοιου είδους πρακτικές για τα θέματα μίσθωσης ε, ή ε, χρήσης ε, τέτοιων αεροσκαφών ώστε να μην λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των εργαζομένων όπως για παράδειγμα πιλότων ή εκείνων που θα είναι υπεύθυνοι για τον χειρισμό τους. Πρέπει λοιπόν από πλευρά ΕΑΣΑ να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά. Αλλά συνολικά με τα όσα αναφέρθηκαν συμφωνώ και σε σχέση με τον κύριο Μίλτενμπεργκ για αυτούς τους τρεις πυλώνες, τους τρεις άξονες ε, και τη σπουδαιότητα των κανόνων και για την ε, υποχρεωτική εφαρμογή αυτών των κανόνων και την υποχρεωτική καταγραφή, καταχώρηση σε μητρό αυτών των αεροσκαφών και τα τέλη που πρέπει να εισπράττονται και στο τέλος αυτά τα αεροσκάφη να μπορούν να σε συγκεκριμένες τεχνικές ρυθμίσεις και περιορισμούς που είναι στοιχεία αναγκαία. Τους, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα συζητήσουμε και θα εξειδικεύσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Φαντάρελ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι άκρος σημαντικό να διαρωτηθούμε πώς θα περιορίσουμε τη γραφειοκρατία τι λύσεις μπορούμε να βρούμε στα προβλήματα που ήδη υπάρχουν από σήμερα ή βλέπουμε να διαφαίνονται για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά την ιδέα όλη αυτή, νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η γνωμοδότηση του κυρίου Μαρινέσκου βασίζονται και οι δύο σε παλιές πολιτικές και αυτό με εκπλήσει. Λένε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Όλο και περισσότερη Ευρώπη. Αυτό λέμε και ξαναλέμε και αυτή είναι η γραμμή που βλέπω. Άρα δεν ξέρω κατά πόσον πρόκειται για τη σωστή προσέγγιση. Εγώ θα έλεγα το αντίθετο. Όπως και αν έχει. Δεν θέλουμε να έχουμε μια αντίδραση που Παυλόφ στην ε, ανάγκη επίλυση προβλημάτων, δηλαδή να απαντάμε ανακλαστικά περισσότερη Ευρώπη χρειάζεται, Ξέρουμε ότι υπήρξε αυτό το ατύχημα, την προηγούμενη εβδομή υπήρξε το δυστύχημα με την ε, πτήση της ε, Egypt. Είχαμε και άλλα ε, με ουκρανικά προβλήματα, με ουκρανικό αεροσκάφος κτλ. Έχουμε τώρα το νέο πρόβλημα με τα drones, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξει μια συντριβή, μπορεί να υπάρξει κάποια σύγκρουση ενό μη επανδρομένου με ένα επανδρομένο και φυσικά απέφχομαι κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να συμβεί μια μέρα. Τα drones μπορεί να γίνουν ένα επικίνδυνο παιχνίδι και να οδηγήσουν σε καταστροφές ή σε καταστροφή. Ο οργανισμό χρειάζεται και νέα εργαλεία, αλλά το κυριότερο που απαιτείται είναι η αύξηση τη ευαισθητοποίηση ε, των χρηστών των drones, των χειριστών αυτών των ε, σκαφών, για να ξέρουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε γιατί πολλοί δεν αντιλαμβάνονται ε, ακριβώς τους κινδύνους. Και σίγουρα αυτό θα πρέπει να συνδέσει με την επιβολή της νομοθεσίας. χρειαζόμαστε λιγότερη ατιμορρησία. Ακούσαμε για τεχνικούς περιορισμούς, για άδειε και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά σίγουρα, αλλά θα πρέπει να επιβάλλονται και κυρώσεις εκεί που χρειάζεται να είμαστε πιο αυστηροί το να έχουμε λοιπόν οργανισμούς με περισσότερη, ε, πιο διευρυμένη εντολή κτλ. Αυτά πιστεύω ότι είναι απαρχιωμένες απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και δεν είμαι υπέρ. Επίσης πολύ σωστά νομίζω ένας από τους ομιλητές είπε για τα αερόστατα, ε, για την ομοθεσία στην Ευρώπη. ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε κάποιους κανόνες που ήδη έχουμε ε, για τα αερόστατα, να μην ε, επανεφευρίσκουμε δηλαδή κάθε φορά τον τροχό. Αφού υπάρχουν κάποιες διατάξεις μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ντομινίκ και τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου και εμένα κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του, να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για την πρότασή της. Το S στον ΕΑΖΑ, το safety, σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και στην όλη συζήτηση. Θέλω να υπογραμμίσω το εξή. Στι διεθνεί συζητήσει, όπω διαθρώνονται αυτή τη στιγμή, ιδίω όταν αφορά την πιστοποίηση, δεν έχουμε ε, μία θέση έτσι αρκετά άνετη για τον ΕΑΖΑ απέναντι στους ισοδύναμους αμερικανικό-κινέζικο οργανισμό. Και νομίζω ότι αυτό το έχω πει και επαναλάβει και ο διευθυντής ε, του οργανισμού. Θα ήταν πολύ επωφελές για τον κλάδο ο ΕΑΖΑ να έχει ένα διεθνές καθεστώς ώστε να μπορεί να συνομιλεί ε, ε, ισότιμα με τους ομολόγους οργανισμούς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την υπεράσπιση του κλάδου μας, της βιομηχανίας μας. Άκουσα τον Πέτερ Βαντάλ με πολύ ενδιαφέρον πρέπει να πω μιλά για ευρωπαϊκά ε, παυλόβια αντανακλαστικά, αλλά υπάρχουν και τα εθνικιστικά, τα λαϊκιστικά αντανακλαστικά πάλι τύπου Παυλόφ. Και θα έλεγα ότι αυτή η δραστηριότητα εξορισμού ε, θα μπορούσε δύσκολα να γίνει αντικείμενο ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο μόνο, νομίζω. Ποιο είναι όμως το πραγματικό ζήτημα. Είναι παράδοξο να γίνεται λόγος. Έχουμε εδώ ε, πάλι το, την αντίδραση Παυλόφ ε, στα, περί Μιλάμε για μείωση του διοικητικού φόρτου, την απλούστευση της νομοθεσία να γίνει πιο αποτελεσματική ε, και να έχουμε μία νομοθεσία και όχι 28 διαφορετικές. Όλα αυτά ε, τα καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία. Εδώ όμως, με τα drones, έχουμε ένα αναδυόμενο πρόβλημα. Υπάρχουν χώρες που μπορούν να αντιδράσουν πολύ πιο γρήγορα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γιατί σίγουρα κανείς μπορεί να τα βρει πιο εύκολα στη χώρα του παρά με 28, 27. Και κάποιες χώρες σίγουρα μπορούν να ρυθμίσουν τα πράγματα, αλλά εκκαινώντας από διαφορετικέ αφετηρίες ενδεχομένως. Όμως τα drones πετάνε παντού, όχι πάνω από μια χώρα μόνο ή μια περιοχή συγκεκριμένη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, έχουμε μια νέα βιομηχανία που αναδύεται ε, και θέλουμε να δούμε και τι θα κατασκευάσει η βιομηχανία, θα τα διαθέσει αυτά στο εμπόριο και ποιοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν. Και ούτε σίγουρα θέλουμε να επιβάλλουμε ένα κατανόητο διοικητικό άρθρο στις χώρες. Θυμάστε με τα κινητά τηλέφωνα. θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε κάθε χώρα να έχει τις δικές της ρυθμίσεις. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με 28 διαφορετικές νομοθεσίες στην κινητή τηλεφωνία, άρα καλό είναι ίσως να μην επαναλάβουμε το ίδιο λάθος. Όπως είπε και ο Μάτιε τώρα, ε, σίγουρα όσο περισσότερο ε, αυξάνουμε το φόρτο εργασίας αλλά μειώνουμε ε, τον προπολογισμό του οργανισμού, ε, και το βλέπουμε πολλές φορές, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον οργανισμό να κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά, ιδίως για ένα τόσο σημαντικό ε, θέμα. Και με ξενίζει πολύ περισσότερο που και η Κομισιόν ε, δεν θέλει να ρυθμίσει προϋπολογισμούς που δεν δίνει τελικά όπως σημαίνει το συγκεκριμένο οργανισμό, γιατί τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού δεν προέρχονται από τα κοινοτικά ταμεία. Να ρυθμίσει το δέχομαι κατά κάποιο τρόπο το δικό της ε, μερίδιο η Κομισιόν, αλλά να ρυθμίζει έναν προπολογισμό που δεν, στον οποίο δεν συνεισφέρει ή τέλο πάντων συνεισφέρει μόνο εν μέρη, κάπως με ξενίζει. Ευχαριστώ. Ε, Μαρή Κριστίν Νοτιού, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Μαρινέσκο και τους ε, διάφορους εισηγητές τους οποίους άκουσα προσεκτικά. Πολύ γρήγορα. Να χαιρετήσω καταρχάς το έργο του ΕΑΣΑ, που είναι πολύ σημαντικό και είναι και διεθνώς αναγνωρισμένο. Αλλά ομολογώ ότι έχω μπερδευτεί λίγο για την εξέλιξη του οργανισμού. Αυτή η σταδιακή προέκταση της εντολής του ε, μπερδεύεται λίγο με τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών, ε, της ε, ΙΑΣΑ και του Eurocontrol. έχουμε κινδύνους πραγματικούς ε, επικαλύψεων, ε, δημιουργίες ε, διοικητικών αχθών που θα ήταν προβληματικά για τον ευρωπαϊκό κλάδο αεροπλοείας και αθέμητο ανταγωνισμού επίσης. Εγώ θα επιθυμούσα ο οργανισμός να επικεντρωθεί στο ρόλο του που είναι ρόλος στήριξης των εθνικών αρχών και συντονισμού σχετικά με τις διατάξεις ασφαλείας που προέρχονται από την Τώρα, σχετικά με τη συζήτηση που διεξήχθηκε στην Ιταλική Γερουσία, ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία που ε, προκύπτουν κάποια στοιχεία που δεν σέβονται ακριβώς την επικουρικότητα. Ε, ναι, κύριε Ρικέ, και για τη χώρα μας έχει σημασία αυτό. Και αυτό ισχύει και για τις υπηρεσίες εδάφους και για τα αεροσκάφη, για την πιστοποίηση, για την αδειοδότηση και για το πεδίο εφαρμογής των ε, κατευσιώτησης πράξεων, για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις εθνικές αρχές ε, προς τον ΕΑΣΑ, τα κράτη-μέλη, λέει ο εισηγητής, μπορούν να αποκαταστήσουν τις αρμοδιότητες ε, που είχαν απολέσει λόγω ασφαλείας, όταν αυτό δεν αφορά σε συγκεκριμένες ελλείψεις βεβαίως. Όμως, είναι σημαντικό οποιαδήποτε διάταξη ασφαλείας να γίνει σε απόλυτη συνεργασία με την ΙΑΣΑ και με διατάξεις που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα μπορούσαν να εκτιμήσουν ως υπερβολικά αυστηρούς ή περιοριστικούς. Χρειαζόμαστε μια προσέγγιση που να προστατεύσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου αεροπλογίας και θα προτείνουμε κάποιες ε, τροπολογίες προς την κατένση αυτή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σβάκ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης ε, και την Επιτροπή και τα όσα έκανε ο κύριος Μαρινέσκου για την έκθεση αυτή. Ένα ζήτημα με απασχόλει και είναι η μετάθεση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών εναντί της ΕΑΣΑ. Η ερώτησή μου ουσιαστικά είναι αυτό θα σημαίνει μετάθεση αρμοδιοτήτων επίσης και από την Ευρωκοντρόλ προς την ΕΑΣΑ τέτοιων αρμοδιοτήτων. Υπάρχει μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Eurocontrol και η ερώτησή μου αν η απάντηση είναι καταφατική είναι ναι ότι οι αρμοδιότητες από την ε, Eurocontrol θα μετατεθούν στην ΕΑΣΑ θα θέλω να γνωρίζω αν αυτό αφορά την απόφαση του Συμβουλίου Δεκεμβρίου 2015 και συνάδει με αυτήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις από πλευρά μου. Καταρχάς και το άρθρο 32 που αφορά στις ε, πρόσθετες υπηρεσίες εδάφους και τα σλότ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εδώ το κείμενο που λέγει ότι θα πρέπει να κατεδεικνύεται ότι υπάρχει η απαραίτητη δυνατότητα για το δυναμικό. Δεύτερον, τα μία επανδρομένα δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει αύξηση της χρησιμοποίησης των drones. Και επομένω, πριν την ανάπτυξη της αγοράς αυτής θα πρέπει να έχουμε ήδη τοποθετήσει απαραίτητα στοιχεία ασφαλείας. Επομένως θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχει ε, πολύ συγκεκριμένη και αποτελεσματική εξέταση των πιστοποιητικών και των αδειών, αλλά εδώ ε, το ζήτημα έχει και διασυνοριακή διάσταση και επομένως ε, αυτό αφορά την επιχειρησιακή δυνατότητα και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών των διαφόρων φορέων. Θα χρειαστεί και αυξημένη ασφάλεια σχετικά με τις αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τις εθνικές αρχές προς τον οργανισμό και τέλος, μία παρατήρηση, ενδεχομένως έχουμε μία υπερβολική ποσότητα κατεξιοδότηση πράξεων, γιατί ναι, δεν μπορούμε να επιβαρύνουμε πάρα πολύ το διατακτικό, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι θα παρέμβομαι επί πολύ ουσιαστικών. Με περιορισμένη επομένως δυνατότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων να μπορούν να παρεμβαίνουν στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ζήνε παρακαλώ έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Μαρινέσκου, λέει η κυρία Μάισνερ, για την έκθεσή του. Τρει ε, επί τη αρχή παρατηρήσει ε, για το θέμα και ε, όσον αφορά και τι τροπολογίε επίση. Το ένα και εμένα με απασχολεί το θέμα του συσχετισμού ΕΑΣΑ Eurocontrol. Υπάρχει ο προβληματισμό να υπάρχει στην Ευρώπη μια αρχή που θα είναι αντίστοιχη εκείνη στον ΗΠΑ. Όμω, το να πούμε ναι εντάξει με το Eurocontrol έχουμε πολλές αρμοδιότητες που λειτουργήσε η υπηρεσία σωστά και εγώ θα έλεγα ότι και αναφέρθηκε και από αρκετούς η δομή θα έπρεπε να διατηρηθεί και φυσικά θα πρέπει να έχει περαιτέρω αρμοδιότητες η ΆΣΑ σωστό αυτό να το σκεφτούμε αλλά χρειάζονται και οι δύο στο μέλλον και θα ήθελα ως δεύτερο σημείο να δούμε ότι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα εναντί των εθνικών ρυθμίσεων. Έχουμε ευρωπαϊκούς εθέρες και πρέπει να υπάρξει αυτός ο ευρωπαϊκός χώρος στη ρύθμισή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι λοιπόν και οι δύο οργανώσεις πρέπει να επιμεριστούν το έργο τους και να έχουν καλή συνεργασία μεταξύ τους. Το άλλο αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Από πλευρά ε, συναδέλφου αναφέρθηκαν οι τρεις αρχές. Ε, εντάξει σίγουρα χρειαζόμαστε κανόνες και Εκεί όπου έχω κάποιες επιφυλάξεις ή σκέπτομαι κάποια θέματα ε, σε σχέση με φιλελεύθερες ε, πρωτοβουλίες για παράδειγμα, να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τους ιδιωτικούς ε, τέτοιους επιχειρηματίες μη επανδρομένων αεροσκαφών. Το να δούμε το αν θα μπορούν να, δεν θα μπορούν να υπερβούν κάποια όρια, κάποια σύνορα. Εντάξει, αλλά να δούμε και το θέμα των χειρισμών και ελιγμών. Δεν ξέρω πώς τεχνικά μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά, θα έπρεπε να μην ε, υπαρισφρέουμε στην ε, ιδιωτική δραστηριότητα υπερβολικά και επιβαρύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία. Εντάξει, και για τα καθήκοντα ρύθμισης και διαχωρισμού, διαφοροποίησης αυτών πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε καλύτερα. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να οδηγήσει να έχει προτεραιότητα η ασφάλεια να και να είναι λειτουργικές οι προτάσεις. Και το άλλο θα δω όλες τις προτάσεις ε, προσεκτικά. Ξέρω ότι στις ΗΠΑ για παράδειγμα καλύτερα από εμά εδώ στην Ευρώπη ρυθμίζεται το πώς τα τεχνικά συστήματα ε, για για την αναγνώριση αεροσκαφών σε σχέση με, τις μεγάλες, ε, με τα μεγάλα αεροσκάφη διαφοροποιούνται. Πρέπει εδώ να δούμε σε σχέση με τους εθέρες ε, με το, την ε, ΕΑΣΕ να έχουμε ένα σύστημα που θα διασφαλίζει αυτές τις πτυχές ασφάλειας. Δεν είναι δυνατόν μεγάλες, μεγάλα αεροσκάφη να έχουν διαφορετικό εξοπλισμό από μικρά και να έχουν έτσι διαφορετικές δυνατότητες ταυτοποίησης και εντοπισμού των άλλων αεροσκαφών. Αυτά πρέπει να ρυθμίσουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ντανιέλα Αγιούτο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για τον Ιασά εμείς ανησυχούμε ε, σχετικά με αυτήν την περσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων στον οργανισμό. Με τι πόρους θα γίνουν αυτά αφενός. Αφετέρου θα έχει την απαραίτητη δυνατότητα ο οργανισμός να αναλάβει όλες αυτές τις εντολές και αρμοδιότητες. Επίσης ο σχετισμός ε, μεταξύ ΕΑΣΑ και Eurocontrol. Η μεταφορά κάποιων αρμοδιοτήτων θα μπορούσε να δημιουργήσει σύγχυση και συγκρούσεις. Συγκρούσεις για παράδειγμα, ε, όσον αφορά τη διαμόρφωση τελών. Εμείς ε, πρέπει να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση εξέβρεση λύσεων περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Θα πρέπει δηλαδή να επιβραβεύονται κάποια σύντομα δρομολόγια, πιο μικρά, τα οποία όμως έχουν μεγαλύτερο κόστος. Χρειάζεται επίσης να συζητήσουμε τις συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων, των εργαζομένων και τις συνθήκες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού πτήσεως. Γιατί υπάρχουν κάποια σκοτεινά σημεία σχετικά με τις υφιστάμενες παρούσες συνθήκες ε, συμβάσεων για τους ε, εργαζομένους αυτούς. Επίσης δεν μας πείθει ε, ο σχετισμός των διατάξεων ασφαλείας με την επίδοση. Τώρα όσον αφορά στη συζήτηση των μη επανδρομένων είμαστε υπέρ απολύτως του να δούμε το θέμα αυτό στο κείμενο με εστίαση επί της ασφάλειας και επί της προστασίας ιδιωτικότητας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εγώ ίδιο έχω μια σύντομη παρατήρηση ολοκληρώνοντας. Η κυρία Τζακί Φώστερ αναφέρθηκε στις Delegated Acts ε, όταν αναφέρονται τέτοιε πράξει γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θέλουν μέσω αυτής της διαδικασίας να αποφασίζουν αποκλειστικά για λογαριασμό του τι θα γίνεται. Κάθε φορά έχουμε αυτή τη συζήτηση για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξη, ε, πράξης. Ε, μας ανακοινώνονται, έχουμε τρεις μήνες περίοδο για να πούμε ότι εντάξει ωραία, μπορούν να γίνουν τεχνικά αυτά, να ρυθμίζονται έτσι ή θέλουμε να εμπλεκόμαστε εμείς. Εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να αποφασίζουν και να, λένε, να λέμε ότι είναι πολιτικά τα θέματα αυτά και δεν μπορούμε εμείς να εξαιρούμεθα. Κάθε φορά όταν έχουμε τέτοιου είδους τριμερών διαλόγων delegated εντάξει, είναι εξαιρετικό μέσο να εξοικονομούμε χρόνο, αλλά είναι και ένα μέσο να αποκλείεται το Ευρωκοινοβούλιο και να μην συμμετέχει. Δική μας δουλειά είναι να πούμε και να λέμε αυτά είναι τεχνικά θέματα, στα άλλα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουμε. Δεν γίνεται κάθε φορά να ξαναξεκινάμε όλα αυτά από μηδενικό σημείο. Έχει ε, δέκα χρόνια τώρα η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Είναι σαφή πλέον τα πράγματα. Ως κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι πρέπει να προσέξουμε να μην ακολουθήσουμε τέτοιου είδου παιχνίδια παιχνίδια και να λέμε ότι εντάξει ωραία χαιρόμαστε να μην συμμετέχουμε και εμπλεκόμεθα. Έχουμε λίγο χρόνο για κάποιες ε, ε, δηλώσεις. Ε, δεν είχα αντιληφθεί ότι πρόκειται για μία άμεση ερώτηση. Θα θέλαμε λοιπόν να δούμε πώς αυτό θα μπορέσει να ρυθμιστεί. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια ερώτηση. Ωραία. Ο κύριος εισηγητής... Α, όχι, μια στιγμή. Προηγούμενα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά, φυσικά Πώς μπορούσα σε σχέση με αυτά τα, τις, αυτές τις κατεξουσιοδότηση πράξη να αφήσω εκτός την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθόλου. Εδώ λοιπόν εμπλέκεστε, έχετε τον λόγο παρακαλώ Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με λυπεί που μας ε, θυμηθήκατε μόνο στο πλαίσιο των κατεξουσιοδότηση παράξεων. Ελπίζω να υπάρχουν και πιο θετικά, ε, συνενετικά πράγματα που μας ενώνουν. Τέλος πάντων, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Μαρινέσκου για το σχέδιο έκθεσης. Γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλο, μακροσκελές το κείμενο της πρότασης, ε, το διήλθε, το διέτρεξε διεξωτικό τρόπο και διατύπωσε και μια δέσμη προτάσεων Πολλές από τις τροπολογίες του έχουν στόχο να ενισχύσουν ε, το σύστημα της Ευρωπαϊκής Αεροπορίας, την ασφάλεια, να ενισχύσουν τον ΕΑΖΑ και όλα αυτά εν είναι ευπρόσδεκτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μας ικανοποιεί επίσης ε, το ότι ο βασικός ή μάλλον οι βασικοί στόχοι της πρότασης Κομισιόν ε, υποστηρίζονται από τον εισηγητή Μαρινέσκου και αν, τολμώ να πω και αυτό ε, συνάγω από τη συζήτηση που άκουσα σήμερα. Ο στόχος του κειμένου είναι η μετάβαση προς ε, ένα περιβάλλον που θα βασίζεται περισσότερο στις επιδόσεις ε, και σε πολιτικές σχεδιασμένες βάσει των κινδύνων. Θέλουμε επίσης οι αλλαγές που θα επιφέρουμε να μας επιτρέψουν να κάνουμε πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο. Τρίτον, θέλουμε να καλύψουμε κάποια κενά τα οποία φάνηκε ότι έχει το ρυθμιστικό σύστημα, το ground handling, η ασφάλεια. Και τέλος, στόχος μας είναι καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν να αντιμετωπίσουμε τις αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν μεταξύ της ασφάλειας της αεροπλοείας και άλλων ε, τομέων που επηρεάζουν, έχουν τεχνικό αντίκτυπο, όπως είναι η ασφάλεια της αεροπορίας και η υπερστασία του περιβάλλοντος. Θέλουμε να βελτιώσουμε το κείμενο ως προς αυτές τις πτυχές και το ανέφεραν και πολλοί ευρωβουλευτές σήμερα το πρωί στις παρεμβάσεις τους. Έρχομαι τώρα σε κάποιες πιο συγκεκριμένες απαντήσεις για το τελευταίο ζήτημα αυτών των αλληλεξαρτήσεων. Στον τομέα της ασφάλειας ε, θα έχετε παρατηρήσει ότι ο στόχος μας δεν ήταν να διευρύνουμε ε, το πεδίο αρμοδιοτήτων του ΕΑΖΑ, γιατί δεν είναι ένας ε, οργανισμός ασφάλισης από την έννοια του security, αλλά ένας οργανισμός ασφάλισης από την έννοια του safety, προστασίας. Και ε, αυτό που θέλουμε ε, είναι να ρυθμίσουμε καλύτερα τα πράγματα για να λάβουμε υπόψη αυτές τις αλληλεξαρτήσεις. Κάτι που αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, ως παράδειγμα, είναι αυτές οι εμπολίμες περιοχές, οι περιοχές συγκρούσεων. Εκεί ε, αυτές οι δύο πτυχές της ασφάλειας, safety και security, ε, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Και μετά από συζήτηση στο Συμβούλιο, έχει ενισχυθεί και το κείμενο σε αυτό το σκέλος του. Ελπίζω το στήριξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης τώρα, περιβάλλον, εδώ τονίζουμε αυτές τις αλεξαρτήσεις, ε, ώστε να λαμβάνονται πλήρως υπόψη από τον ΕΑΖΑ. Δόθηκε ένα παράδειγμα δηλαδή ότι έχουμε πιο ελαφρύ αεροσκάφη για εξοικονόμηση καυσίμου. Φυσικά, η χρήση νέων υλικών ε, πρέπει να συνοδεύεται και από εξασφάλιση ότι είναι ασφαλή τα υλικά αυτά. Ο ΕΑΖΑ θα πρέπει όμω να λαμβάνει υπόψη και την πτυχή τη ασφάλεια και την πτυχή όμω ε, των περιβαλλοντικών ε, ωφελών από πιο ελαφρά αεροσκάφη. πολύ επίση ανέφεραν θα πρέπει ε, να υπάρξει στενή διασύνδεση με τα πρότυπα τη ΔΟΠΑ και συμφωνούμε. Το ίδιο ισχύει και για τα πρότυπα ασφαλεία. Αυτό που ωστόσο προτείνουμε να αλλάξει σε σχέση με τον εφιστάμενο κανονισμό είναι αυτόματη ένα προς ένα αντιγραφή των περιβαλλοντικών προτύπων ε, του ΙΚΑΟ. Δεν το έχουμε αυτό στην ασφάλεια. Προτείνουμε να εφαρμοστεί στο περιβαλλοντικό σκέλος ό,τι ισχύει για την ασφάλεια. Δηλαδή, απριόρι στηρίζουμε και οθετούμε τα πρότυπα ε, του ΙΚΑΟ, της ΔΟΠΑ. Όχι όμως ένα προς ένα. Δεν το κάνει και κανείς άλλο στον κόσμο. Αυτό νομίζω ότι αποδυναμώνει και τη διαπραγματευτική μας θέση στο πλαίσιο της ΔΟΠΑ για να έχουμε το καλύτερο δυνατό περιβαλλοντικό, ε, τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά πρότυπα. Έχουμε στο Eurocontrol και τη σχέση με τον ΕΑΖΑ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι δεν αλλάζουμε, ούτε καν προτείνουμε αλλαγή στα αρμοδιότητε ή ευθύνε του ΕΑΖΑ σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τη ενέργεια κυκλοφορίας Αυτό έγινε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν από αρκετά χρόνια, συγκεκριμένα το 2009. Ο ΕΑΖΑ ανέλαβε κάποια καθήκοντα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείριση, τα drones, ε, ναι, κυκλοφορία και άρχισε να εκπληρώνει αυτά τα νέα καθήκοντα. Αληθεύει ότι προέκυψαν κάποια ζητήματα, κάποιες αλληλεπικαλύψεις με το Eurocontrol. Αυτό είναι φυσιολογικό γιατί είμαστε σε μεταβατική περίοδο και πρέπει να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα που μιλάμε υπάρχει μια ομάδα εργασίας με Eurocontrol, ΕΑΖΑ και Κομισιόν ε, που επεξεργάζεται ένα κατάλογο ε, επιμερισμού των αρμοδιοτήτων, ώστε ο καθένας να ξέρει ποια είναι τα καθήκοντά του, η εντολή του και να μην υπάρχει αλληλεπικάλυψη ε, και σε ό,τι αφορά ε, το ανθρώπινο δυναμικό. Ελπίζουμε να έχουμε ολοκληρώσει αυτό το κατάλογο μέχρι το καλοκαίρι. Σε ό,τι αφορά αυτές τις, αυτά τα τέλη για τα οποία αναφέρθηκαν, στα οποία αναφέρθηκαν κάποιοι, εμείς θέλουμε εν μέρη ο ΕΑΖΑ να χρηματοδοτείται όταν μιλάμε για το ATM, Τέλο πάντων να υποφελείται από αυτέ τα, τα οδικά τέλη, root charges που καταβάλει η βιομηχανία, Όπω ισχύει για οποιονδήποτε δραστηριοποιείται στη διαχείριση ανέργεια κυκλοφορία, εθνικέ αρχέ, Eurocontrol, οτιδήποτε έχει να κάνει με ATM, διαχείριση ανέργεια ε, το διαχειριζόμαστε μέσω αυτών των τελών. Αυτό που δεν γίνεται όμω είναι ε, η εποπτική, ε, ο υποπτικό ρόλος. Δεν λαμβάνεται υπόψη τα ATM. Ουσιαστικά λοιπόν ε, ακολουθούμε τη λογική που ισχύει εδώ και χρόνια στο ATM. Και επίσης προσθέτουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά δεν θα υπάρξει συγκεκριμένα ε, μεταφορά ε, κονδυλίων. Θα αλλάξει νομοθεσία για το σύστημα έσπρεξη αυτών των τελών απλά και μόνο. Για να υπάρχει μια δυνητική μεταφορά των τελών αυτών στον ΝΕΑΣ. Δεν το επιβάλλουμε όμως, το προτείνουμε. Και βέβαια αν θα γίνει κατά τρόπον ώστε να μην αυξάνει το συνολικό κόστος των χρηστών των αερίου χώρου, δηλαδή των αεροπορικών εταιριών. Γιατί σε περίπτωση αυτή θα ε, μιλάμε για μετατόπιση κάποιου, μετακύληση ε, κάποιου τέλους και δεν μιλάμε για προσθήκη ενός νέου τέλους. Άρα δεν θα επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος, ούτε οι χρήστες του εναέρου χώρου. Τελευταίο σημείο. Drones. Airman Έτσι είναι όρος. Αναδιόμενος ο τομέας, το είπατε κι εσείς. Υπάρχει συνένεση σαφής, πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε. Έχουμε την ευκαιρία να δράσουμε σωστά, επειδή ξεκινάμε από το μηδέν. Και πρέπει να σας πω ότι μετά από ένα-δύο χρόνια συζητήσεων και με την έκθεση της κυρίας Μπόστο, υπάρχει νομίζω όλο και μεγαλύτερη συνένεση ως προς το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ασφάλεια των drones, να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας ε, αυτού του τομέα να αναπτυχθεί και της ασφάλειας και των ανθρώπων που βρίσκονται ε, στο έδαφος ε, και την ασφάλεια στον αέρα. Σε αυτή τη φάση το ερώτημα είναι, σε αυτόν τον κανονισμό, πόσο, σε ποιο βαθμό πρέπει να ασχοληθούμε. Εγώ θα έλεγα να μην βάλουμε σε αυτόν τον κανονισμό όλες τις λεπτομέρειες, γιατί δεν το κάνουμε ούτε για άλλους τομείς της ασφάλειας αεροπορίας για τα σκανισμού ε, για την αεροπλοημότητα. Δεν το κάνουμε αυτό. Δεν λέμε πόσες ε, ε, θύρες εξόδου, πόσες θύρες εξόδου emergency exit θα πρέπει να έχει ένα αεροσκάφος. Δεν πάμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Το ίδιο λέμε και για τα drones. Να βάλουμε κάποιες βασικές απαιτήσεις. Η πρόταση είναι στο παράρτημα και να συμπεριλάβουμε κάποιους διαδικαστικούς κανόνες όπως κάνουμε και σε άλλους τομείς και να μείνουμε εκεί. Γνωρίζω ότι είναι εύκολο ο πειρασμό να προσθεθούν λεπτομέρειε. Γιατί φυσικά οι λεπτομεριακοί κανόνε που αναπτύξει ε, δεν υπάρχουν ακόμη, δεν του βλέπουμε. Δώστε μα όμω, σα παρακαλώ, χρόνο για να αναπτύξουμε αυτού του αναλυτικού λεπτομεριακού κανόνε και α παραμείνουμε εδώ ε, σε κάποια γενικά καθήκοντα. Διότι στο μέλλον θα αλλάξει η τεχνολογία και εμεί θα έχουμε κολλήσει με κανόνε που δεν θα μπορούμε να προσαρμόσουμε. Ένα τελευταίο σχόλιο. Η εντύπωσή μας και το επιβεβαιώνει νομίζω και η σημερινή συζήτηση, είναι ότι δεν πρόκειται για μια άκρο επίμαχη νομοθεσία. Υπάρχει ευρία συνένεση επί πολλών πτυχών φυσικά και θα υπάρξουν τροπολογίε. Πρέπει να πω όμω ότι βλέπω και σημαντικέ βελτιώσει για τον τομέα ε, τη ε, αεροπορία Και οι βιομηχανία και οι εθνικές είναι κάτι που το περίμεναν για να μπορούν να γίνουν προσαρμογές και στους αναλυτικού κανόνες. Άρα, έκκληση που απευθύνω είναι και ελπίζω να έχουμε οριστικοποιήσει και εγκρίνει αυτόν τον κανονισμό ε, σύντομα, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές και να εγκρίνουμε για παράδειγμα του αναλυτικούς κανόνες για την ασφάλεια των drones. Αυτή είναι η έκκλησή μου λοιπόν. Ευχαριστώ και εδώ ολοκληρώνω. Ευχαριστώ και για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ. Και πρωτού δώσω και πάλι τον λόγο στον εισηγητή. Θέλω να διορθώσω αυτό που είπα. Η συνθήκη της Λισαβόνας το 2010, έξι χρόνια έχει ηλικία και όχι δέκα, έκανα λάθος. Και τώρα ο κύριος Μαριάν Μαρινέσκου έχει τον λόγο παρακαλώ. Thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάποια σχόλια πρώτα όσον αφορά τα θέματα αυτά για την, ε, τις αρμοδιότητες ε, αυτής της αρχής ε, και σε σχέση με τον τίτλο της. Καθώς θεωρώ ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την έκθεση της κυρίας Φώστερ που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο όσον αφορά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την έκθεση για τις τροποποιήσεις της ε, ΕΑΣΑ από και τις τροποποιήσεις του ιδίου του Κοινοβουλίου ήταν νομοθετικού χαρακτήρα αυτή η νομοθετική έκθεση όπου δεχθήκαμε και εγκρίναμε να έχουμε μία εθνική αρχή μόνο αρμόδια, όχι πολλές ε, διαφορετικές και που άλλαξε ο τίτλος ε, αυτός ε, όσον αφορά το όνομα. Γιατί, για διάφορους λόγους, ε, αερο, αερομεταφορές συνεπάγονται ασφάλεια. Δεν μπορεί να λειτουργούν χωρίς ένα πελαίσιο ασφάλειας. Όταν έχουμε λοιπόν χάρη της ασφαλείας την ευρωπαϊκή αυτή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών, όσον αφορά της, το δεύτερο επίπεδο, επιβάλαμε αυτό το δεύτερο επίπεδο το 2009 όταν θεσπίσαμε μέσω των ρυθμίσεων την Εθνική Εποπτική Αρχή. Και τώρα κάποια χρόνια μετά μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε μία αρχή πλέον και για πολλούς διαφορετικούς λόγους και για λόγους χρηματοοικονομικούς, προϋπολισμού κτλ για την ε, κοινωνική ασφάλεια έχω εισαγάγει μια, έχω καταθέσει μια τροπολογία σε σχέση με αυτό που εντάσσεται ήδη στον κανονισμό και νομίζω ότι επαρκεί για τα αεροδρόμια να υπάρχει μια εξαίρεση, θα μπορούσε να είναι μια εξαίρεση όσον αφορά τα μικρά αεροδρόμια αλλά τα περισσότερα αεροδρόμια θα υφίστανται αυτή τη ρύθμιση. Όσον αφορά την Eurocontrol, τέλη, ίσπραξη, τελών, και σύγκρουση συμφερόντων. Εγώ από ό,τι πιστεύω σήμερα μπορούμε να κάνουμε λόγο για σύγκρουση συμφερόντων. Και αυτό γιατί, διότι λαμβάνει χρήματα από τέλη διαδρομών η Eurocontrol και ταυτόχρονα δρά ως ε, ρυθμιστική λειτουργική αρχή που αφορά τα θέματα τα λειτουργικά όσον αφορά την θέσπιση ε, τελών διαδρομών. Αυτό επιλύεται μέσω του κανονισμού που εμείς ψηφίσαμε κατά το παρελθόν, όπου εμείς ζητήσαμε τα PR, δηλαδή τα θέματα αποτελεσματικότητας, πρέπει να καλύπτονται από έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό φορέα. Εγώ εισήγαγα λοιπόν επίσης ε, και μια τροπολογία ώστε να διαχωριστούν οι αρμοδιότητες, να αποσαφινιστούν τουλάχιστον οι αρμοδιότητες, να μην υπάρξουν διπλοεπικαλύψεις μεταξύ Eurocontrol και EASA. Και πιστεύω επίσης ότι αυτό επαρκεί. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για όλα τα σχόλια και παρατηρήσεις σας. Θα τα λάβω σίγουρα υπόψη για την σύνταξη και κατάθεση τροπολογιών. Ευχαριστώ επίσης τους επαΐοντες που παρέστησαν και μας προσφώνησαν. Πρόεδρε, αν έχουμε χρόνο μπορώ να θέσω ένα ερώτημα προς τους επαΐοντες. Έχουμε άλλα 9 λεπτά μια πολύ σύντομη απάντηση θα μπορούσε να δοθεί στο ερώτημά μου. Λοιπόν, η ερώτησή μου λοιπόν είναι, είσαστε ικανοποιημένοι με τις κατηγορίες αυτές που προτείνονται από την ΕΑΣΑ σε σχέση με την ΕΑΣΑ στην τεχνική γνωμοδότηση, τεχνικού χαρακτήρα γνωμοδότηση και ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τις δύο κατηγορίες ε, όσον αφορά τις ε, ε, αυλαβής πτήσης με σαφή κριτήρια και με βάση σαφή τεκμήρια και την άλλη κατηγορία όλων των άλλων περιπτώσεων. Σας ικανοποιεί αυτή η ρύθμιση. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε λοιπόν τώρα παρακαλώ να παρέμβει. Εσείς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Όπως εξήγησα, η βασική μας ανησυχία είναι με την ανοιχτή κατηγορία. Θα θέλαμε να έχουμε μια κατηγορία χαμηλού κινδύνου, όπως χειριζόμαστε σε άλλα πεδία, όπως τα παιχνίδια, και μία άλλη που σχετίζεται με την αεροπλοεία και τις διατάξεις ασφαλείας χαμηλού κινδύνου της αεροπλοείας. Αεροπλοείας, με συγχωρείτε. Η ανοιχτή κατηγορία, ως έχει αυτή τη στιγμή, και καθότι δεν έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία, από ό,τι δηλαδή καταλαβαίνουμε μέχρι τώρα δίνει την εντύπωση πολύ υψηλότερου κινδύνου από αυτά που λένε αυτοί που προωθούν το κείμενο. Μάλιστα σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 8 Ιουνίου 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ και πάλι τους πραγματονόμονες, και προσβλέπω σε ε, ότι ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση και για σας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης τώρα. So we have to continue. Συνεχίσουμε λοιπόν, καθίστε ή αποχωρήστε αν δεν επιθυμείτε να παραμείνετε. Περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Ησυχία παρακαλώ. Είναι η βελτίωση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας των μεταφορο... μεταφορικών υποδομών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη ήθελα όσοι δεν επιθυμείτε να αποχωρήσετε γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις μας. Ή καθίστε παρακαλώ. Εντάξει. noch einmal. Λοιπόν, και πάλι η βελτίωση των συνδέσεων και της προσβασιμότητας μεταφορικών υποδομών στην Κεντροανατολική Ευρώπη. Η συγητής είναι ο Τόμας Πιότρο Πορέμπα. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, συνάδελφοι. Πολύ χαίρομαι που σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησής μου, έκθεσης, σχετικά με την βελτίωση των συνδέσεων και της προσβασιμότητας των ε, μεταφορικών υποδομών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Και η γνωμοδότηση αυτή θα έπρεπε να καταστεί ένα από τα κεντρικά στοιχεία, τα πιο σημαντικά στοιχεία της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής μεταφορών για τα επόμενα χρόνια, θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Πιστεύω πως σήμερα μπορούμε να πούμε ότι επί τη βάση των όσων ήδη έχουμε αποφασίσει με τα TNT και τις ε, ε, Connecting Europe Facility σχετικά με την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ε, υποδομές μεταφορών και έως ε, τα μέσα της δεκαετίας του 2020 έχουμε ήδη ε, καταρτήσει ένα πλαίσιο και είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε πιο σημαντικά προβλήματα και πιο συγκεκριμένα προκλήσεις που σχετίζονται με την βελτίωση της διασυνδεσιμότητες μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαιτέρως των κρατών μελών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πολωνία, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Και να σας αναφέρω ένα-δύο στοιχεία σχετικά με τα βασικά προβλήματα συνδεσιμότητας που αντιμετωπίζουμε στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα είναι μια έλλειψη συνοχής, συνάφειας αν θέλετε, ε, οικονομικός και εδαφικός μιλώντας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις συνδέσεις λοιπόν των περιοχών και των κρατών αυτών και κυρίως αναφέρομαι στα έργα που σχετίζονται με τα αισθήματα μεταφορών τα οποία θα πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικά θα πρέπει να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να προσελκύσουν επενδύσεις. και νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει και ένα πλαίσιο ευκαιριών ε, περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ανάπτυξης σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης. Αλλά πώς πρέπει να αντιλαμβάνεται κανείς την καλύτερη συνδεσιμότητα και την καλύτερη προσβασιμότητα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, των οδικών δηλαδή και των συνδυνομικών μεταφορών αλλά και των αεροπορικών των αερομεταφορών. είναι ένα στοιχείο που θα μας επιτρέψει να προστατεύσουμε καλύτερα και τα ανατολικά μας σύνορα και συνολικά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας από τους πυλώνους που διασφαλίζουν ε, την προστασία και την ασφάλεια των κρατών μελών είναι οι κρίσιμες υποδομές μεταφορών σε όλο το μήκος, αν θέλετε, των ανατολικών συνόρων, όλο και πιο σημαντικό θέμα σήμερα. Νομίζω ότι οι επενδύσεις σε αυτές τις κρίσιμες υποδομές θα μπορούσαν να ε, σημαίνουν, να μεταφραστούν σε καλύτερη ασφάλεια για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη συνολικά. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω την αναγκαιότητα της ανάπτυξης καλύτερων και ευρύτερων συνδέσεων σε αυτό το τμήμα της Ευρώπης. Περισσότερες ανατολικές περιοχές θα μπορούσαν να γίνουν τμήμα του δικτύου τέντη. Αυτό θα οδηγούσε σε δυνατότητες ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης. Αυτά τα βήματα είναι πολύ σημαντικά και ήδη τα βλέπουμε σε έργα όπως το έργο των Βαλτικών Σιδηροδρόμων και εδώ θα ήθελα να χαιρετήσω τις δεσμεύσεις και της Κομισιόν και των ενεχομένων κρατών μελών. Εκτιμούμε επίσης την αποφασιστικότητα της νέας πολωνικής κυβέρνησης που θεωρεί το Rail Baltica ως ένα από τα βασικότερα προγράμματα, έργα για τις μεταφορές για τα επόμενα χρόνια. Οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνουν περισσότερα ώστε να εκμεταλλευτούμε το ήδη φυστάμενο πλαίσιο, αυτά που ήδη έχουμε επιτύχει. Κάποιες διαβουλεύσεις έχουν ήδη λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια, την Κομισιόν. Υπάρχει και ένα άλλο έργο που αξίζει μία στο Βία Καρπάτια από τη Λιθουανία ως την Ελλάδα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένας πολύ σημαντικός άξονας οδικός που θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη για όλες τις χώρες που διατρέχει από τη Βαλτική ως τη Μεσόγειο αλλά είναι ένας άξονας οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου που θα μπορούσε να σημαίνει και καλύτερη και αυξημένη ασφάλεια των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και συνολικά, λέει ο μιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επενδύσεις ε, στις υποδομές αυτές σημαίνουν και πόρους και νομίζω ότι και η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να συντονιστούν καλύτερα. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί απόλυτη συνέπεια σε όλες τις δράσεις και πρωτοβουλίες που θα αναλυθούν, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου είδους μεταφοράς και θα πρέπει να εξασφαλιστούν επίσης να επιτευχθούν συνέργειες και στη χρηματοδότηση. Μεταξύ της διευκόλυνσης Connecting Europe, της ε, Τράπεζας Επενδύσεων, και της καλύτερης χρησιμοποίησης των υφιστάμενων πόρων ή στο πλαίσιο των κονδυλίων για τις ε, στρατηγικές επενδύσεις. Όλα αυτά θα μας βοηθούσαν να υλοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά έργα υποδομών μεταφορών σε αυτές τις ευρωπαϊκές περιοχές. Επίσης η μακροπεριφερειακή συνεργασία και η χρησιμοποίηση μηχανισμών καινοτομίας διακυβέρνησης. ώστε να επιληθούν προβλήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση και τις μεταφορές που δεν μπορούν τα κρατημέλη από μόνο τους να επιλύσουν. Και υπάρχουν συσχετισμοί ευρεία στρατηγικής για όλες τις σχετιζόμενες περιοχές, τη Βαλτική, το Αιγαίο, το Ιόνιο, την περιοχή των Καρπαθίων και ο δικό άξονας της Βία Καρπάτη οπωσδήποτε θα ήταν η ραχοκοκαλιά αυτή της μελλοντική ε, στρατηγική. Για τις ε, χερσαίε υδάτινε ή αέρες μεταφορές, η αεριε μεταφορε η εκθεση μας οπωσδήποτε θα πρέπει να εστιαστεί στην προώθηση των συνδέσεων μεταξύ ειδών μεταφοράς πρέπει να επιτύχουμε περισσότερα, να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο στις συνδέσεις της υλοδρομικές, γιατί είναι σαφές ότι σε αυτό το μήμα της Ευρώπης δεν είναι όσο ανεπτυγμένες θα έπρεπε. Και για τους επιβάτες και για τα εμπορεύματα. Και τα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα αυτή και να βελτιώσουν την κατάσταση στα επόμενα χρόνια. Δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί επαρκής οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών χωρίς επαρκής επενδύσεις στον τομέα αυτών. Κάτι ακόμα που ήθελα να αναφέρω στην εκθεσή μου και ελπίζω να μπορέσετε να το υποστηρίξετε είναι η χρησιμοποίηση του δυναμικού τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπης εις ό,τι αφορά στι εσωτερικέ υδάτινε μεταφορέ, τις εσωτερικέ πλωτέ οδούς όπως ο Δούναβη, που είναι πολύ σημαντικοί άξονες. Θα πρέπει οι σχετικέ χώρες να εξασφαλίσουν καλύτερη χρησιμοποίηση των πλωτών αυτών οδών. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούμε απολύτως αποτελεσματικά τις εσωτερικές πλευρές οδούς, τους ποταμούς, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε Πολωνία, Τσεχική Δημοκρατία και Αυστρία μέσω των οδών αυτών με πολύ καλύτερο τρόπο και στη Βαλτική και στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλύτερα τους λιμένες και στη χρησιμοποίηση ε, των ενεργειακών πόρων, αλλά και στα θέματα ασφαλείας. Επίσης, οι εγκαταστάσεις στον πυθμένα της θάλασσας δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες των λιμένων, ούτε να είναι εμπόδιο πως προς συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουμε στους ε, λιμένες εισόδου. Και εδώ αναφέρομαι συγκεκριμένα στο έργο Nord Stream, που δεν είναι απόλυτα εποφελές σχετικά με την προσβασιμότητα συγκεκριμένων λιμένων συμπεριλαμβανομένων σημαντικών λιμένων στην Πολωνία. Συνάδελφοι, ω εισηγητή, θα ήθελα να σα ε, διαβεβαιώσω ότι είμαι απολύτω ανεκτός σε προτάσεις και σε περαιτέρω συζήτηση για να βελτιώσουμε περαιτέρω την έκθεση. Νομίζω ότι η συνδεσιμότητα και η προσβασιμότητα της ε, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι πάρα πολύ σημαντική. Ελπίζω να ακούσω ενδιαφέρουσες ε, προτάσεις και σκέψεις και από εσά. Θα πρέπει να συνεργαστούμε υπό την βασική αρχή και κατεύθυνση ότι το κείμενο αυτό θα πρέπει να καταστεί ένα κείμενο που θα συμπεριλαμβάνει στρατηγικές κατευθύνσεις που θα μας βοηθήσουν, θα μας βοηθήσουν για το μέλλον να βελτιώσουμε την συνδεσιμότητα και την προσβασιμότητα στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη ως στρατηγική προτεραιότητα. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στην έκθεση κάποιες διατάξεις επί τη βάση των οποίων το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα στο μέλλον στο πλαίσιο οποιοδήποτε έργου για τις μεταφορές που θα μπορούσε να έχει εποφελείς λύσεις και εξέλιξη για τις περιοχές αυτής της Ευρώπης. Δεν μιλούμε μόνο για την προσβασιμότητα των μεταφορών και τις καλύτερε συνδέσεις. Δεν είναι μόνο για την κάλυψη ενός κενού οικονομικής ανάπτυξης ή μιας εστέρησης. Δεν είναι απλώς για την η επιτάχυνση της οικονομικής μεγεθύνσης της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά είναι η προστασία και η ασφάλεια του συνόλου του εδάφους Ευρωπαϊκής Ένωσης. οι αποτελεσματικέ ε, μεταφορικές συνδέσει σε όλα τα είδη μεταφορών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι στην πραγματικότητα η δυνατότητα αύξησης της αίσθησης ασφαλείας των κατοίκων των περιοχών αυτών αλλά και συνολικά όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι κάτι που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μία από τις βασικές κατευθύνσεις, από τα βασικά μηνύματα που θα πρέπει να διαβιβάζονται από το κείμενο αυτό και από τις θέσεις της Επιτροπής μας. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα μπορέσετε να συμφωνήσετε με τις προτάσεις μου και όπως έλεγα περιμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τη συνεργασία μαζί σας για να αναπτύξουμε περαιτέρω το κείμενο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα να συγχαρώ τον κύριο Πορέμπα η έκθεσή του πιστεύω ότι είναι εξαιρετική βάση για το έργο που πρέπει να καλύψουμε και όπως προαναγγέλθηκε θα είναι λέει ανοιχτός, με ανοιχτό πνεύμα θα αντιμετωπίσει προτάσεις τροπολογιών και εμείς από πλευρά του ΕΛΚ θα καταθέσουμε τέτοιες ε, τροπολογίες και κυρίως ε, εκείνο το οποίο θέλουμε να καλωσορίσουμε είναι το ότι αυτή η πρόταση μπόρεσε να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη των εργασιών μας αυτό το θέμα. Και κατά τα άλλα ελπίζουμε ότι η έκθεση αυτή θα δώσει κίνητρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει και θα κινητοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τις εργασίες της επ' αυτού. Είναι μια πρόταση λοιπόν πόσον αφορά την έκθεση αυτή τη θεωρούμε πολύ θετική. Είναι πολύ θετικό το ότι η έκθεση αυτή καλύπτει τον οριζόντιο τρόπο προσανατολισμού και προσέγγισης εγκάρσια. Είναι μια πολύ σημαντική πτυχή αυτή η συνιστόσα. Και είναι και πολύ σημαντικό από την άλλη πλευρά να δούμε και τον βορρά-νότο ως άξονα, να ενδυναμωθεί ο άξονας βορρά-νότου στις διασυνδέσεις αυτές, ώστε τα ε, εμπλεκόμενα κράτη-μέλη να πρέπει και από πλευρά τους να μεριμνήσουν για τα σύνορα και τις διασυνδέσεις. Και θα διαδραματίσει αυτό και υστερότερα, μεταγενέστερα, ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικά και η προσπελασιμότητα, η προσβασιμότητα όσον αφορά τις διασυνδέσεις ε, πρέπει να αναφέρεται και να διασφαλίζεται διότι έχει επιπτώσεις στα κράτη-μέλη και στις όμορες, στις γειτονικές χώρες και ούτως ή άλλως όπως στη Λευκορωσία, Μπελαρούσια παράδειγμα. Αλλά αφορά επίσης και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων οπωσδήποτε. Τώρα υπάρχουν, υπάρχει και ένας πολύ σημαντικός ρόλος σε αυτά τα ανατολικά σύνορα. Η ανάπτυξη των υποδομών, η ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών μπορούν να έχουν όλα αυτά θετικές επιπτώσεις ε, στις ε, προαναφερθήσεις όμορες χώρες και να έχει θετική επίπτωση αυτό στην οικονομική τους ανάπτυξη μέσω αυτών των διασυνδέσεων. Και επιπλέον μπορεί να ε, συνεισφέρει και στην πολιτική σταθεροποίηση των χωρών αυτών. Κάτι άλλο τώρα. Έχουμε και περαιτέρω προτάσεις, ιδέες, πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε συνέχεια ώστε να μπορέσει να εμπλουτιστεί και να ε, μετεξελιχθεί αυτό το κείμενο. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τους μηχανισμούς χρηματοδότησης για παράδειγμα, προγράμματα υποδομών, είναι πολύ σημαντική η χρηματοδότηση ως συνιστόσα Εχθές ακούσαμε από την Επίτροπο κυρία Μπούλτς όσον αφορά τις χώρες συνοχής για παράδειγμα, συγκεκριμένες προτάσεις και έχουμε πολλά να μάθουμε επ' αυτού και πολλά να κάνουμε, να πράξουμε. Εξάλλου θα πρέπει να οδηγηθούμε και στην κατάθεση τροπολογιών και να διαβιβαστούν στον εισηγητή και ευελπιστούμε στο ανοιχτό πνεύμα ώστε να γίνουν δεκτές οι προτάσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Κλάουδια Ταπάντερ έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την δουλειά που έκανε στα πλαίσια της ακτής αυτής ε, και εμείς ε, από πλευράς ε, ομάδας σοσιαλιστών έχουμε μια θετική προσέγγιση εδώ και συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει αυτή η πρωτοβουλία να συζητηθεί διεξοδικά στην Επιτροπή Μεταφορών. Και περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον και την παρέμβαση της Κομισιόν. Αυτό το κείμενο καλύπτει όλα τα στοιχεία που είναι τα πιο σημαντικά για την ανάπτυξη των υποδομών στις μεταφορές. Είναι ισορροπημένο, χειρίζεται ισορροπημένα και σωστά τις διαφορές μεταξύ των περιοχών, μας προετοιμάζει για το μέλλον. Σε ό,τι αφορά στις προτεραιότητες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι σαφές ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας των μεταφορών και θα πρέπει να ανακτήσουμε ε, και το κοινό που μας χωρίζει από την ε, Δυτική Ευρώπη σε αυτό το επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ένα μεσοπρόθεσμο ε, πρόγραμμα αναπτυξιακό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις περιοχές και θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να συνεργαστούν οι εθνικές αρχές με τις ενωσιακές. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας αυτής, ιδιαίτερα για τα πιο ουσιαστικά στοιχεία του προγράμματος. Θα πρέπει να έχουμε συνεργασία στις στρατηγικές επιπαραδείγματι της μακροπεριφερειακής συνεργασίας, της ανταλλαγής ε, ε, αρμοδιοτήτων, της ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών, αλλά όλα αυτά θα εξαρτηθούν και από τους συμμετέχοντες και από τον προϋπολογισμό. Αν δεν υπάρχει συνεργασία όλων των ενεχομένων φορέων δεν θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα στοιχεία αυτά. Επίσης οι διασυνδεσιμότητες μεταξύ διαφόρων ειδών μεταφορών, μεταξύ για παράδειγμα των σιδηροδρομικών συστημάτων, των πλωτών οδών, του οδικού δικτύου, είναι πολύ σημαντικές. Κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό σε εμπορικό επίπεδο είναι η, η διαφορετική χρησιμοποίηση των μέσων μεταφοράς, αλλά πάνω απ' όλα και θα ήθελα να το υπογραμμίσω οι εμπορικοί και οι οικονομικοί φορείς χρειάζονται ευελιξία ώστε να επιλέξουν το καλύτερο σύστημα μεταφοράς. Αυτό που τους εξυπηρετεί καλύτερα ακόμα και αν επιθυμούν να περάσουν από ένα σύστημα σε ένα άλλο. Να θυμίσω επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο για τα κρατημέλη να διαχειρίζονται πολύ συχνά τα συστήματα ιστορικών πλωτών οδών. Αναφερθήκατε στο Δούναβι. Εμείς έχουμε ήδη δύο συμφωνίες επ' αυτού που υπεγράφησαν από τις ε, ενεχόμενες χώρες, από τα κράτη και αυτό είναι πολύ σημαντικό πιστεύω. Έχουμε τις ε, δεσμεύσεις του Ρότερνταμ. Ελπίζω τα κράτη-μέλη να σεβαστούν αυτές τις δεσμεύσεις. Για εμάς ο Δούναβης είναι ο άξονα σύνδεσης μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Έχει μια τεράστια εμπορική οικονομική σημασία, αλλά έχει και τεράστιο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ποτάμι που καταλήγει στο ποτάμι της Κωνσταντσίας στη Μαύρη Θάλασσα να αναπτυχθεί αλλά σε συνεργασία και σε ισορροπία με το Ρότερνταμ ακριβώς για να αναπτυχθεί αυτή η συνέργεια μεταξύ Δύσεως και Ανατολής. Για μας είναι θεμελιωδέστατο. Βεβαίω και υπάρχουν διάφορα συστήματα μεταφορών τα οποία συγκλίνουν αν θέλετε με τον άξονα του Δούναβη για τη συνδέση με τις υπόλοιπες ε, περιοχές της Ευρώπης. Αλλά αυτά τα έργα υποδομών τόσο μεγάλης κλίμακος για τις μεταφορές Χρειάζονται στήριξη από τα ευρωπαϊκά ταμεία και κονδύλια. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες οι χρηματοδοτικέ δυνατότητες που υπάρχουν και θα πρέπει να συμμετάσχει και ο ιδιωτικό φορέας μέσω συμφωνιών ιδιωτικού δημοσίου. Όμως, πάντοτε αντιμετωπίζουμε, όπως λέμε, προβλήματα χρηματοδοτικά, προβλήματα που οφείλονται πολύ συχνά στο συντονισμό που απαιτείται εσωτερικά στα κράτη-μέλη με μια σειρά αρμοδίων φορέων με τους οποίους πρέπει να συνεργαστεί κανείς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις διασυνδέσεις ε, προς την ε, κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι η απλούστευση της διαδικασίας ε, αδειοδότησης για έργα υποδομών μεταφορών. Είναι απολύτως απαραίτητη αυτή η απλούστευση, επίγει θα έλεγα, πάρα πολύ συχνά είναι εξαιρετικά επαχθής και μακροσκελής αυτή η διαδικασία. Πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν συγκεκριμένα τι έχει γίνει επ' αυτού, ποια είναι η πρόοδος που έχει σημωθεί σε κάθε κράτος. Αυτό είναι απαραίτητο εάν θέλουμε να προσαρμοστούμε λίγο περισσότερο προς τις ευρωαϊκές απαιτήσει για τις πτυχές τις εξωτερικές. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι είναι απαραίτητο να εξετάσουμε τις ε, δυνατότητες διασυνδέσεων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους άμεσους γείτονες, με τα όμορα κράτη τα τρίτα. Αυτό είναι ουσιοδέστατο για τις εμπορικές μας σχέσεις, για τις οικονομικές μας σχέσεις η βελτίωση για παράδειγμα των συνδέσεων με τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία που είναι περιοχέ πολύ σημαντικέ για την οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα τη Ευρωπαϊκή Υπήρου λέει ο Μιλήτρια. Θα πρέπει όμως επίσης να δούμε πώς θα συνδεθούμε με τις βασικούς άξονες ε, μεταφορές του Καυκάσου για παράδειγμα και για τη μεταφορά εμπορευμάτων από και προς την Κίνα όπως και περιοχές για τις οποίες, ε, επί των οποίων αυτή τη στιγμή υφίστανται κυρώσεις ή περιορισμοί. Θα πρέπει να ξαναδούμε όλη τη στρατηγική μας για το Δυτικό Κάφκασο, μαζί με τα θέματα ενέργειας, μεταφορών και στρατηγικής πολιτικής. Και αυτά άπτονται και ε, του τουρισμού, που είναι απολύτως απαραίτητο κομμάτι της οικονομίας για πάρα πολλές ευρωπαϊκές περιοχές. Καθότι αναπτύσσουμε δίκτυα υποδομών μεταφορικών, θα πρέπει να αντίστοιχα να αναπτύξουμε δίκτυα τουριστικών υποδομών. Υπάρχουν πάρα πολλές πολυεθνικές εταιρείες που θέτουν περιορισμούς ή μάλλον προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συστημάτων τοπικής εμβέλειας σε κάποιες περιπτώσεις. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες ζώνες, ποιες περιοχές ε, μου λείπει, έχω ακόμα ένα λεπτό, λέει η ομιλητρία πρόεδρε, μιλώντα πάρα πολύ γρήγορα. Ε, εν πάση εμεί έχουμε τεράστιο δυναμικό στην Ευρώπη τουριστικό, αλλά δεν μπορούμε απλώ να υπολογίζουμε πάνω στην συνδεσιμότητα και την ε, προσβασιμότητα. Θα πρέπει να βρούμε και άλλε λύσει και άλλε διεξόδου, ώστε να φτάσουμε στι ε, περιοχέ ε, των κρατών μα που είναι ο τουρισμό πιο σημαντικό. Το τελευταίο θέμα που θέλω να αναφέρω είναι ο χώρος ε, Σέγγεν. Είναι σαφές ότι εδώ συζητούμε περισσότερο στο πλαίσιο των υποδομών, αλλά οι υποδομές είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωαϊκής κινητικότητος. Και τελευταίος, κάποιες χώρες ε, θέτουν εμπόδια αντί να τα έρουν. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία, στη Βουλγαρία με συγχωρείτε, ε, κοιτάξτε, λέει ο Πρόεδρο, το, το λεπτό σα ε, ξεπεράστηκε. Αν όλοι ε, οι ομιλητές είναι τόσο μακροσελεί, δεν θα τα καταφέρουμε. Ε, δηλαδή, εντάξει, έχετε αναφερθεί και στο Σέγγεν, στη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική, ας εστιαστούμε λίγο. Ναι, ήθελα όμως, Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μία φράση για να κλείσω. Ε, καθότι είμαι και σκιώδης ε, εισηγήτρια φαντάστηκα ότι θα μπορούσα να αναπτύξω κάπως περισσότερο την απόψή μου φαντάστηκα πρόεδρε θα πρέπει λοιπόν αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας να είναι να παρέχει ε, ένα καλό feedback, μια σωστή ανάλυση και πλήρη ανάλυση σχετικά με όλες τις πτυχές που σχετίζονται με το πρόβλημα της ανάπτυξης μιας επαρκούς ε, ε, δομής, υποδομής μεταφορών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη που πρέπει να σχετίζεται με τη στρατηγική TNT. Θα πρέπει να υπάρχει η χρηματοδοτική στήριξη διότι αλλιώς δεν θα επιτύχουμε τίποτα. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε ένα, μια ανάπτυξη που να είναι ενσωματωμένη και ισορροπημένη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως, ισορροπημένη δηλαδή οικονομική ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Αλλά δυστυχώς Πρέπει να πω ότι περιορισμό ε, στις παρεμβάσεις ε, σε, πέντε λεπτά πρέπει να θεσπιστεί, διαφορετικά δεν μπορέσουμε να τα βγάλουμε. Ευχαριστώ. Μπορώ όμω ίσως σύντομα να πω και εγώ κάτι, λέει η κυρία Μάισνερ, Μία παρατήρηση ήθελα μόνο να κάνω, διότι και ο Δούναβης φυσικά βρίσκεται ιδιαίτερα στο επίκεντρο και για την τελευταία περίοδο πάντα αναφερόταν η διασύνδεση από τον Ατλαντικό μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα αυτή και η πρόταση αυτή για μια διοργάνωση είναι σημαντική να δούμε αν υπάρχει μια δυνατότητα να ακολουθηθεί. Ευχαριστώ. Εντάξει, ευχαριστώ. Εσεί τώρα έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να παραστώ κατά τη διάρκεια τη παρουσίαση από πλευρά του εισηγητή. Υπήρχαν ε, αλληλοσυγκρουόμενε ε, συνεδριάσει ε, και στι υποχρεώσει μου όσον αφορά την έκθεση. Πρέπει να πω ότι δεν είμαι ιδιαίτερος, ιδιαίτερα οπαδό μια έκθεση που συγκεκριμένα θα αναφέρεται μόνο σε ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με κάποια αναφορά, αλλά όμως ε, αυτό ε, πρέπει να μας κάνει να ενδιαφερόμαστε για την κεντροανατολική Ευρώπη σφαιρικά. Υπάρχουν πολλά εδώ τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά ταυτόχρονα όπως και στη Δυτική Ευρώπη είναι γεγονός ότι οι κεντροανατολικές ευρωπαϊκές χώρες δεν χρησιμοποίησαν πάντα, όπως και η δική μου, με αποτελεσματικό τρόπο τα κονδύλια που διέθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για διάφορους λόγους. Δεν είμαστε προετοιμασμένοι, δεν υπήρχαν προγράμματα, δεν υπήρχαν μελέτες επιπτώσεως περιβαλλοντικές πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές τα κονδύλια τα οποία ε, χρησιμοποιήθηκαν ε, πολλές φορές ε, συνεπαγόντουσαν υψηλότερες, υψηλότερη δαπάνη. Δεν βρίσκω ιδιαίτερα να επικεντρώνεται το σχέδιο έκθεσης στην ασφάλεια, σε σφαιρικά στις πτυχές της ασφάλειας. Και αυτό είναι κάτι που με τις τροπολογίες που κατέθεσα προσπάθησα να αποκαταστήσω ως ισορροπία είναι έκθεση βέβαια για την κεντροανατολική Ευρώπη, αλλά κυρίως φαίνεται ότι είναι μια αναφορά στην Ανατολική Ευρώπη, στις Βαλτικές χώρες, στην Πολωνία, στις χώρες με τα ανατολικά σύνορα. Η κεντρική Ευρώπη κάπως εδώ δεν ε, εντάσσεται ε, ως αντιστάθμισμα. Και αν δει κανείς ε, τη διασύνδεση βορρά-νότου-ανατολής-δύσης, θα πρέπει λοιπόν να αναφερθούμε σε αυτό το περίπλοκο πλαίσιο. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω, η Βιολέτα Μπούλτσα αναφέρθηκε χθε εδώ, μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις για το μείγμα πολιτικών ή τις, ε, ε, τις διάφορες, ε, τους διάφορους συνδυασμούς. Αλλά πρέπει να δούμε και τις συνέργειες, να μην υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα αλλά αλληλοσυμπληρούμενα έργα και προγράμματα. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε στην προσέγγισή μας. Κατανοώ βέβαια την επικέντρωση στις οδικές μεταφορές από πλευράς του. Υπάρχει όμως και κάποια μη σώροπη σχέση εδώ με ισχυρή επικέντρωση στους δρόμους, στις οδικές μεταφορές και όχι τόσο στους σιδηροδρόμους η αναφορά περιβαλλοντικά. Εντάξει, να μπορέσουμε να αναφερθούμε στις ανάγκες που πρέπει να, να καλύψουμε, οι τροπολογίες μου θα αποκαταστήσουν ε, την ισορροπία μεταξύ διαφορετικών τρόπων ε, μεταφορών ε, οδικών και σιδηροδρομικών. Τώρα στρέφομαι στα κονδύλια, στη χρηματοδότηση. Κάνει λόγο ο εισηγητής για έναν ε, θεμητό έντιμο ανταγωνισμό και τις ανάγκες και τις ε, ε, ιδιομορφίες των κρατών μελών. Αυτό που πρέπει να μεριμνήσουμε είναι να επανεισάξουμε ή να ξαναδούμε το ευρωπαϊκό σύστημα το, το οποίο θα ισχύει στο μέλλον όποιο και αν εγκριθεί και θα προαχθεί είναι κάτι το οποίο θέλω να προτείνω να εντάσσεται με πιο ολοκληρωμένο τρόπο στο μέλλον από ό,τι μέχρι σήμερα. Ολοκληρώνω πρόεδρε. Πράγματι θεωρώ ότι δεν πρέπει να επισέλθω σε όλα τα σχόλια τα οποία ε, θα γίνουν μέσω των τροπολογιών μου. Αυτό που θέλω να κάνω είναι κάποιες ε, μη σχέσεις να αντισταθμιστούν, να εξισορροπηθούν και να, εισαγάγω κάποια, να εισαχθούν κάποια στοιχεία, μια και κάνουμε λόγο για την κεντροανατολική Ευρώπη, την δημοκρατία της Τσεχίας για παράδειγμα δεν αναφέρονται κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Αναφέρεται ο Δούναβης, αναφέρονται οι βαλτικές χώρες, δεν αναφέρονται όμως ε, συγκεκριμένοι διάδρομοι που θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν. Όλα αυτά σε σχέση με μια σταθερή βάση ως θεμέλιο για να εργαστούμε θα εισαγάγω τροπολογίες να εξισορροπήσω περισσότερα τα πράγματα για την ασφάλεια σφαιρικά, για τη συμπληρωματικότητα, για τα συστήματα και τη μέθοδο εισπάξης διοδίων και τελών. Θα συνεργαστώ με τον εισηγητή ώστε να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα είναι προς όφελος όλων. Πρόεδρος, ευχαριστώ και έτσι παρακαλώ. Ε, κύριο Σκρέλετς, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πορέμα για την έκθεσή του και πιστεύω ότι αυτό το θέμα και εδώ πρόκειται για ένα σχέδιο έκθεσης είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των συστημάτων μεταφορών, μεταξύ των χωρών που είναι τα περισσότερο ανεπτυγμένα, ε, οι περισσότερο ανεπτυγμένες στην Ευρώπη δυτικές ευρωπαϊκές χώρες και των άλλων που είναι κεντροανατολικοευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε ω θέμα, στη δική μας κοινοβουλευτική επιτροπή και σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές που ασχολούνται με τις πολιτικές χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχή αυτών των, συνοχής αυτών των κρατών. Και θεωρώ εξίσου ότι είναι θεμελιώδους σημασία αυτό το οποίο ε, σχολίασε ο συνάδελφος, ότι επενδύουμε πολλά ποσά και γίνονται πολλές προσπάθειες για τους σιδηροδρόμους. Η απουσία υποδομών στις ε, κεντροανατολικοευρωπαϊκές χώρες έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μεταφορά αγαθών αλλά και επιβατών σε σχέση με τις χώρες αυτές. Και κάτι ακόμα, επιπλέον οδηγεί στο σε σχέση με τις μεταφορές μας να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές ρήπων μέχρι το 2030, εκπομπές που θα προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών. Πρέπει να αναπτύξουμε συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών ταμείων που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη και μέσω προϋποθέσεων και κριτηρίων που θα αντανακλώνται μέσω της νομοθεσίας με τον μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα μετατρέπονται σε βιώσιμα προγράμματα και σχέδια μακροπρόθεσμα. Πρέπει επίσης να πετύχουμε μια καλύτερη διασύνδεση και καλύτερη προσβασιμότητα στις υποδομές μεταφορών αυτών των περιφερειών και περιοχών. Αλλά πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλους στόχους που έχουν και αυτή κεφαλαιώδη σημασία. Μείωση των εκπομπών ρήπων σε αέριες μεταφορές, μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, ε, επίσης το να μπορέσουμε να είμαστε σφαιρικοί κάποιο πιο αποτελεσματική, επιτυγχάνοντας ισότητα των επενδύσεων, ισότιμους όρους για τις επενδύσεις μεταξύ αυτών των χωρών. Και αυτό αφορά και τις υποδομές. Πρέπει επίσης να εναρμονίσουμε τις διατάξεις ώστε να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε τις διαφορετικές περιοχές και περιφέρειες. Έχουμε πολλά παραδείγματα απουσίας διασυνοριακών διασυνδέσεων. Όσον αφορά τις επενδύσεις μας θα πρέπει να μπορέσουμε να πετύχουμε πιο αποτελεσματικά και λιγότερο δαπανηρές μεταφορέ. Θα ήθελα επίσης στην έκθεσή σας μια και γίνεται λόγος για τις πολυτροπικές μεταφορές στους λιμένες και στους πρωτού λιμένες πτυχή που είναι πολύ σημαντική ο συνιστόσα για την ανάπτυξη των λιμένων και φυσικά και των σιδηροδρόμων επίσης. Πολυτροπικά. Να μην ξεχνάμε ότι οι σιδηρόδρομοι εξυπηρετούν στο να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους λιμένες. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κύριο Πορέμπα που αναφέρει ότι μέσω καλύτερης διασύνδεσης μπορούμε να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε καλύτερα σε μια μακροπεριφερειακή προσέγγιση. Και πέρα από τη την ε, μακροπεριφερειακή ε, προσέγγιση Βαλτικής Ιωνίου πρέπει να δούμε και την ε, μεγαλύτερη περιφερειακή αυτή ενότητα των Άλπαιων και τις ανάγκες που υπάρχουν εκεί. Για να μην επεκταθώ περισσότερο, θεωρώ ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις υποδομές που ήδη υφίστανται και να τις εκμεταλλευτούμε. Χρειαζόμαστε ωστόσο και την αναγκαία διαφάνεια για την ε, εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και περιβαλλοντικά. Ας μην ξεχνάμε την οδηγία για την ε, Natura 2000 και Ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λουκασεύσκα παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και συγχαρητήρια προς εμάς κύριε Σίγητα. Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια εκθεσή που είναι πολύ σημαντική επειδή ε, φυστά την προσοχή μας σε συγκεκριμένα προβλήματα. Εδώ το πρόβλημα είναι τα κενά και η απουσία διασυνδέσεων σε αυτές τις περιοχές της Ευρώπης. Οι υποδομές φυσικά είναι καθοριστικό συντελέστη της ε, παράγοντας. Ε, ωστόσο δεν θα επαρκεί μόνο αυτή η πτυχή για την διασφάλιση της ανάπτυξης. Παρότι πρέπει να διασφαλιστούν οι υποδομές, οδικές, πλωτές, ε, σιδηροδρομικές, πρέπει να διασφαλιστεί και το θετικό κλίμα για τις επενδύσεις από πλευράς επιχειρήσεων. Με ένα ευνοϊκό σύστημα φορολογίας, αλλά και, ένα, και τη δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού επενδυτικού προγράμματος και περιβάλλοντος. Μην το αμελούμε αυτό. Κάνοντα λόγο τώρα για τους διαδρόμους μεταφορών, ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση όταν διασχίζουν αρκετές χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωση, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη που θα εμπλέκονται και οι κυβερνήσει τους θα μπορούν να υπομισθούν ταυτόχρονα ε, την, την προώθηση, την προαγωγή αυτών των ε, διαδρόμων. Εξίσου σημαντικό για την Πολωνία, Δημοκρατία τη Τσεχία και άλλε χώρε. Όταν υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στην Πολωνία για παράδειγμα και ο εισηγητής και εγώ ζούμε στον πυρήνα, στην καρδιά της ε, Πολωνίας και προς την νοτιότερη περιοχή είναι σημαντικό να δούμε και τα θέματα των Καρπαθίων. Κατανοεί η Πολωνία πολλές φορές καλύτερα αυτά τα θέματα όσον αφορά αυτές τις προτεραιότητες. Η συμβατότητα προτεραιοτήτων είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι ε, εκ των όνου κάνευ. Και μια και η προηγούμενη κυβέρνηση της Πολωνίας είχε υποστεί πολλές επικρίσεις από τον ίδιο τον εισηγητή λέγοντας ότι με τους ρυθμούς υλοποιούν η ε, υλοποίηση της Βία Καρπάτια. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό κάτι σε αυτή τη διαδικασία να υπάρχουν, να διασφαλιστούν οι εγκρίσεις ε, η έγκριση που θα έπρεπε να διασφαλιστεί όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα η περιβαλλοντική μελέτη επιπτώσεων. Αυτό καθυστέρησε τα πράγματα κατά το παρελθόν. Όλοι κατανοούμε όσοι ζούμε σε αυτή την περιοχή ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι οποτεδήποτε θα έχουμε κάποια επένδυση που θα χρειάζεται ταχαίως να διασφαλιστεί πρέπει να κατανοήσουμε ταυτόχρονα ότι πολλές διεργασίες και διαδικασίες που παρακολουθούν και συνοδεύουν αυτές τις ε, εξελίξεις πρέπει να διασφαλίζονται στο ενδεδειγμένο πλαίσιο. Για τη Βία Καρπάτια οι εγκρίσεις που πρόσφατα για παράδειγμα επιτεύχθηκαν Τώρα είναι δουλειά πλέον της ε, ε, πολωνικής κυβέρνησης να ασκήσει την επιρροή της και την πίεση που μπορεί να ασκήσει, να συζητήσει και να διαβουλευτεί με άλλες κυβερνήσεις ώστε να υλοποιηθεί αυτός ο διάδρομος, το αυτός ο διάβλος το δυνατό, το δυνατόν ταχύτερα. Και επίσης ε, κάνοντας λόγο για τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Να επιταχύνουμε τις, ε, ε, την προσέλκυση επενδύσεων, την διάθεση και διασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να τύχουν της ε, υποστήριξής μας και έγκρισής μας. Η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η Επιτροπή Τουρισμού και Μεταφορών είναι μία από τις μεγαλύτερες του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι κρίμα ότι έχουμε τόσα λίγα μέλη από τις περιοχές αυτές ε, των ε, εμπλεκόμενων χωρών. Η απουσία τους δεν θα σημαίνει φυσικά ότι δεν θα τύχει της αναγκαίας υποστήριξης η πρόταση αυτή. Και κάτι άλλο γιατί αναφερθήκατε στη μακροπεριφερειακή στρατηγική, μακρο περιφερειακή στρατηγική για την περιοχή των Καρπαθίων. Ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση. Κατά τα όσα είδα εγώ και εκ της πείρας μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε την υπόθεση αυτής της μακροπεριφέρειας της περιοχής των Καρπαθίων και να λέμε ότι όταν θα εκπονείται μια στρατηγική αυτό δεν θα σημαίνει ότι αυτόματα πρόσθετα κονδύλια θα απαιτηθούν και θα πρέπει να διατεθούν για αυτή την ε, στρατηγική που είναι αναγκαία. Η μακροοικονομική στρατηγική μακροπεριφερειών χρειάζεται πολυτροπικούς και πολύμορφους τρόπους διασφάλισης των πτυχών αυτών των στρατηγικών. Ευελπιστώ λοιπόν ότι αυτός ο διάδρομος θα μπορέσει να προχωρήσει και να υλοποιηθεί. Και θα πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι οποιαδήποτε χώρα με τις καλύτερες υποδομές αν είναι κλειστή σε επενδυτές ε, τότε και δεν υπάρχει ένας ασφαλές πλαίσιο φορολογικό ε, θετικό για τις επενδύσεις και επιχειρήσεις, τότε κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία δεδομένης μιας τέτοιας αρνητικής, ε, ε, ενός τέτοιου αρνητικού δεδομένου. Να το θυμόμαστε αυτό. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ. Αυτό το κείμενο και φυσικά τώρα ολοκληρώνω πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω. Πρόεδρε, θα έπρεπε να επικεντρωθούμε ίσω περισσότερο στους σιδηροδρόμους σε αυτό το κείμενο. Επειδή οι σιδηρόδρομοι είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα των μεταφορών, που είναι εποφελής ε, μέθοδος μεταφορών για το περιβάλλον και πρέπει να αναπτυχθούν σιδηρόδρομοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Έχω εγγράψει και εγώ το όνομά μου στον, ε, στον πίνακα αγοριτών. Δόνα, ε, πριν από 30 χρόνια ήταν το μεγαλύτερο όνειρο των Ευρωπαίων ένα όνειρο να μπορούν από το Ρότεντα μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα να μπορούν ε, να, ε, μεταφέρουν τα αγαθά τους. Ε, εκατομμύρια δαπανήθηκαν και ένας σοσιαλδημοκράτης υπουργός μεταφορών είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη ανοσία μετά τον πύργο της Βαβέλ. Γιατί 80% των πρωτών μεταφορών διεξάγονται στο Ρήνο. Ένα μεγάλο πλατή ποταμό με πρόσβαση στον οκεανό ωκεανό. Το όνειρο επέκτασης πάντα ήταν δεδομένο και στη Βαβαρία διατηρείται αυτό το όνειρο. Αλλά και η βαβαρική κυβέρνηση, η μόνη αρμόδια για αυτό το θέμα, το εγκατέλειψε αυτό το όραμα, αυτό το όνειρο. Στην Αυστρία δεν είναι εφικτό αυτό το όνειρο. Είναι πλωτός ο αλλά όχι για, τα, για μεγάλα πλοία, μεγάλου βυθίσματος. Και έτσι λοιπόν οι προγνώσεις ε, για το Rhein-Main ε, Δούναβη όσον αφορά δηλαδή τον Ρήνο, τον Μίνο και τον Δούναβη μέσω των διορίγων η πρόταση αυτή δεν, είναι, ε, δεν μπορεί να στεφτεί με επιτυχία. Ήταν μια καταστροφή που κατάπιε ως μαύρη τρύπα δισεκατομμύρια χωρίς αποτέλεσμα. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πού θα εντάξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια μας τα οποία δεν είναι ε, απεριόριστα, είναι πεπερασμένα και πρέπει να επιλέξουμε. Αναφέρθηκε ότι απουσιάζει η συνεργασία. Τώρα, ε, συμμετέχουν σε αυτή τη συνεργασία Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Κροατία, Σλοβενία και θέλουν το Amber, δηλαδή του και του ηλέκτρου την, ε, το διάδρομο από τη Βαλτική μέχρι την Αδριατική. Δηλαδή από τη Βαλτική ως την Αδριατική, εξαιρετικό παράδειγμα, διατρέχει εννέα χώρες, μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί, τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχής μπορούν να ενταχθούν εκεί, τεράστιο προτέρημα έναντι άλλων χωρών που το ποσοστό αυτό απαιτείται να είναι πολύ ψηλότερο. Τώρα, συνήθαν και συνεργάζονται αυτές οι χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να τοποθετηθεί επ' αυτού ότι είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί αυτή η διασύνδεση μια και διατρέχει ε, όλες αυτές τις χώρες και διασυνδέεται και με τη Βία Μπάλτικα. Από την Αδριατική ως το Ταλίν θα έχουμε μια εξαιρετική διασύνδεση. Είναι ένα καλό παράδειγμα υφιστάμενων διαδρομών. Δεν χρειάζονται εδώ τεράστιες σύραγγες, τεράστιες γέφυρες. Είναι δυνατόν να μπορέσει με την ηλεκτροδότηση να επιτευχθεί. Θα είχαμε μια εξαιρετική διασύνδεση και όχι μόνο το λιμάνι του Κόπερ του Κόμπαριντ θα μπορέσει να συνδεθεί, θα είναι δυνατόν με πέντε λιμένες να συνεργάζεται. Ο ε, πρόεδρος ε, ο Παύλο Κώστα ε, που από πλευράς Βενετίας είπε δεν θέλουμε να παρατηθέμεθα ως λιμένες και να έχουμε σειράξεις ε, να συνεργαστούμε και συνήλθαν πέντε λιμένες. Ένα θετικό παράδειγμα αυτό, μόνο που δεν αξιολογείται επαρκώς θετικά. Να δούμε αυτή τη συνεργασία των λιμένων αυτών με το διάβλο μέσω αυτών των χωρών θα ήταν εξαιρετικό αυτό. Θα με, ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό αν μπορούσε να υποστηριχθεί ή και με τροπολογία να ενταχθεί. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Συνήλθαν οι χώρες αυτές, ε, στοιχημάτισαν υπέρ του σιδηροδρόμου και έτσι λοιπόν ε, οι πλωτές μεταφορές θα μπορούν να συνδέονται. Ολοκληρώνονται εδώ οι συζητήσεις μας. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει την έκθεση του κυρίου Πορέμπα για τις προκλήσεις τη διασύνδεση και προσβασιμότητας των μεταφορικών υποδομών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Πράγματι, μπορεί να υπάρχουν ε, πολλά κοινά σημεία, αλλά εμεί θέλουμε να δούμε τις ιδιαιτερότητες ε, των χωρών τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπης. Ναι, μεν υπάρχουν ε, υποδομές, αλλά δεν ανταποκρίνεται εντελώ ανάγκη η διάφορες τεχνικές παράμετροι. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού θέλουμε να προσφέρουμε και πιο προσαρμοσμένες ε, λύσεις, ε, όχι μόνο μέσω του Πολιτικού Ταμείου και του Κοινού Ταμείου, αλλά και το Συνδέντας Ευρώ περιλαμβάνει πόρους ε, και διευκολύνει και την εφαρμογή σημαντικών έργων ύψης της αξίας, ιδίως στο σιδηρόδρομο ή τις θαλάσσιε ή μεταφορέ. μεταφορές. Όπως υπεγράμμισε χθε η Επιτροπό Μπούλτ στην ακρόαση, το ΣΕΦ έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό. Ήταν πολύ αποτελεσματική και η πρώτη προκήρυξη διαγωνισμού και υπάρχουν ε, σημαντικά ενωσιακά έργα τα οποία έλαβαν χρηματοδότηση και στη χθεσινή ε, πρόσκληση διαγωνισμού ε, τώρα γίνεται η εξέταση των υποψηφιωτήτων. Θεωρούμε ότι και πάλι θα χορηγηθούν σε μεγάλη ευρωπαϊκή προσθέμενης αξίας προγράμματα τα κονδύλια τα σχετικά με στόχο διασυνοριακές συνδέσεις ε, όπως είναι το Rail Baltica, οι βιώσιμες μεταφορές, η επιλεξιμότητα των, των συνδρομικών ε, έργων περιορίστηκε στα τμήματα τα διοσυνοριακά και αυτά πρέπει να ληφθεί υπόψη και για το σχεδιασμό της επόμενης περίοδου προγραμματισμού από το 2021 έως το 2027 και για την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών δίκτυων στο των μεταφορών. Πάντω, ενισχύθηκε ο προγραμματισμό μας και με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές και την ανάπτυξη των ε, βασικών ε, ε, δικτύων και διαδρόμων. Πολλοί διαδρομοί επηρεάζουν άμεσα συγκεκριμένες περιοχές, βαλτική, αδιατρική ή άλλες, κυρίω σχέσεις και συνδέσει βορρα βορρά-νότου. Η Rail Baltica έχει προχωρήσει γιατί υπάρχει πραγματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, σε υπερεθνικό επίπεδο και Ρήνος Δούναβης. Επίσης εδώ θέλουμε να αναπτύξουμε ε, τη λεκάνη του ποτάμου Δούναβη. Από ευρωπαϊκή πλευρά έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ε, που μεταφράζονται σε επιχειρησιακές κατευθύνσεις. Έτσι θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα για να έχουμε ένα σταθερό περιβάλλον μέχρι την αναθεώρηση του 2023. Πρέπει να δοθεί ε, σωστή ε, προτεραιότητα στη χρηματοδότηση ε, και θα προτείνουμε να δοθεί προτεραιότητα στις βιώσιμες ε, μορφές χρηματοδότησης ε, με στόχο και τους στόχους της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, Έχουμε τα νέα χρηματοοικονομικά μέσα του ΣΕΦ. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτά τα ακούσαμε και στη χθεσινή ακρόαση. Είναι σημαντικά. Τέλος, πολλοί είπαν σήμερα το πρωί και συμφωνούμε ότι υπάρχουν συμφορήσεις ε, και προβλήματα σε ό,τι αφορά τις ρυθμιστικές διαδικασίες, ιδίω όταν μιλάμε για πολύπλοκα έργα υποδομών. Η Κομισιόν λοιπόν θέλει να βρει λύση για τον εξορθολογισμό των συμφορήσεων αυτών και για την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών. Καλωσορίζουμε την έκθεση και ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο. Θα επανέλθουμε μαζί σα για τι επόμενε συνεδριάσει, να σα πούμε πώ προχωρούν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Χαράλτ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για όλα τα σχόλια, παρατηρήσεις. Είναι η πρώτη παρουσίαση της εκθεσής μου, το είπα και πριν αυτό, και σίγουρα τις επόμενες εβδομάδες θα συνεργαστούμε όλοι οι συνάδελφοι για να εκπονήσω το τελικό σχέδιο που θέλω να είναι στο δυνατόν ε, συνεπέστερο με τις δικές σας προσδοκίες. Το έγγραφο αυτό, το είπα και πριν, ε, το αντιμετωπίζω σε ένα στρατηγική σημασία έγγραφο για Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα δηλαδή να μπορέσουμε να ορίσουμε στόχους, στόχους για την Ανατολική Ευρώπη αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη, για τον τομέα των μεταφορών. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποιους μηχανισμούς, κάποιες λύσεις για την ε, ενίσχυση και τη βελτίωση των μεταφόρων σε αυτή την πλευρά της Ευρώπης. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντέλη που μου επισήμανε και τον άξονα βορανό του. Πράγματι, καλή η χρονική στιγμή για να επαναπροσδιορίσουμε και αυτόν τον άξονα και τις κατευθύνσεις που παίρνει ε, η το το των μεταφορών. Και η κυρία Ταπαντέλ πολλά σημαντικά είπε. Την ευχαριστώ. Μίλησε για βελτίωση των διαδικασιών. Γιατί σίγουρα πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα και μπλοκάρονται κάποιες επενδύσεις των μεταφορών και στη δική μου χώρα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ιδίως για την Ανατολική Ευρώπη μιλώ. Έφυγε ο συνάδελφος που δεν ξέρω και αν είχε ακούσει και την ε, αρχική μου ε, παρουσίαση, όπου και είπα ότι η έκθεση θεωρεί ότι η ασφάλεια και προστασία είναι ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα για βελτίωση των μεταφορικών υποδομών στην Ευρώπη. Όλα τα σχόλια θα τα αντιμετωπίσω με πολύ επικοδομητικό τρόπο για την υπέρ της ενεργασίας. Άρα και τα δικά του σχόλια θα τα συμπεριλάβω. Κρόιτς ανέφερε τη σημασία της μακροπεριφερειακής στρατηγικής και μίλησε για μακροπεριφερειακή συνεργασία. Πράγματι, Κάθε στρατηγική έχει και βέλτιστες πρακτικές, ένα κώδικα βέλτιστων πρακτικών. Και αυτό ισχύει και για τον τομέα των μεταφορών. Θα πρέπει να αναφέρουμε και να αποφεληθούμε των στρατηγικών αυτών, γιατί έτσι μπορούμε να αποφεληθούμε και της εμπειρίας που έχουμε συλλέξει για την επόμενη που είχε λάβει το λόγο, πρέπει να πω ότι είμαι ο τελευταίος που θα πω για εσωτερικά πολιτικά ζητήματα εδώ. Αφήνω δηλαδή ε, τις λεπτομέρειες για την στρατηγική μας ό,τι αφορά αυτή την Καρπάθια εδώ Είναι γνωστή η προσωπική μου άποψη, πολλά άλλα θα μπορούσαν να είχαν γίνει, αλλά συμφωνώ ότι αν δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων χωρών που διατρέχει αυτός ο άξονας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ίσως και ανέφικτο να ολοκληρωθεί το έργο. Υπάρχει και ένας θεσμικό χαρακτήρας τις τελευταίε εβδομάδε και μήνες. Δηλαδή, υπήρξε μια δήλωση την οποία επέγραψαν οι Υπουργοί Μεταφορών των χωρών τη Καρπαθίας Οντού. Όλε οι χώρες. Υπεγράφει στην Βαρσοβία μάλιστα η συμφωνία ε, κατά πρωτοβουλία της νέας πολωνικής κυβέρνησης. Υπεγράφει πολιτική δήλωση των Υπουργών Μεταφορών. Για τις χώρες αυτές λοιπόν δηλώνεται ότι η ε, κατασκευή αυτού του οδικού άξονα είναι ύψης της σημασίας. Ένα άλλο σημείο που λέγεται είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθεί και η συνεργασία μεταξύ των χωρών για την ανέγερση αυτού του, για την οικοδόμηση αυτού του δικτύου. Είναι σημαντικό να υπάρχει πολιτική βούληση και να είναι και εμφανής. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο, που πολύ σωστά είπε ότι η συνεργασία μεταξύ χωρών σε ό,τι αφορά και τι ε, θαλάσσιες μεταφορές είναι πάρα πολύ σημαντική. και πρέπει να υπάρχει συνέπεια και με τη λογική με γνώμη την οποία κινούμαστε στον τομέα των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέτοια έργα πάντα θα στηρίζονται από Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν στο πλαίσιο των αναλαμβανόμενων δράσεων, αν υπάρχει αυτή δηλαδή η προσέγγιση. Θα δω λοιπόν τις πρωτοβουλίες αυτές που μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα και μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη των μεταφορών στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις αδρομικές μεταφορές θέλω να τονίσω για μια ακόμη φορά ότι αν θεωρούμε ότι δεν έχει δοθεί επαρκής έμφαση στις σιδηροδρομικές μεταφορές μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Όμως εγώ θεωρώ ότι οι σιδηροδρομικοί και οι σιδηροδρομικές υποδομές είναι σημείο κλειδί για την ανάπτυξη των χώρων. Αν δεν υπάρχει ένα καλό σιδηροδρομικό δίκτυο, Καμία χώρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο με τη Rail Πιστεύω θα προχωρήσει αυτό το έργο και θα υπάρχει ξυπρόδος. Δεν ξέρω, ίσως την εκθέσή μου, ίσως θα μπορούσα να το τονίσω περισσότερο το σκέλος αυτό της διασύνδεσης της σιδηροδρομικής. Θα προσπαθήσω. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή συνάντηση. Σας ευχαριστώ που ε, είχαμε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψε για το σχέδιο εκθεσή μου. Όλοι θα είμαστε ε, συντάκτες αυτού του κειμένου και θα βοηθήσουμε όλοι να βελτιωθούν οι υποδομές των μεταφορών στην Ανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πρόθεσμια κατάθεση τροπολογιών. Δευτέρα Ιουνίου 18.00. Ολοκληρώθηκε η πρωινή μα συνεδρίαση. Στις 3 θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας.